Uh, Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Όπω είπα και χτε, θα το ξεκινήσουμε 9 ακριβώ. Βέβαια, μην νομίζετε, επειδή δείχνει το ρολόι 9 και 7, πάει μπροστά. Έχουμε απαρτία. Ε, Σα καλωσορίζω πρώτα απ' όλα στη συνεδρίαση. Οι συντονιστέ συναντήθηκαν χθε. και πήρε τα πρακτικά τη συνεδρία των συντονιστών. Αν έχετε σχόλια, κύριος Κάζα. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτό που είπαμε και στους συντονιστές. Ήθελα να αναφερθώ στο εξή. Νομίζω ότι κατά τι συνεδρίε των συντονιστών αποφασίσαμε σχετικά με τις επισκέψεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδυάσουμε την επίσκεψη στην Ιαπωνία με μια επίσκεψη στην Ταϊβάν. Αλλά αυτό δεν αναφέρεται σε πρακτικά, γι' αυτό σας λέω ε, να σας ζητώ να μου διευκρινίσετε το σημείο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Κάζαρ που το αναφέρατε. Έχετε πολύ το δίκιο. Η απόφαση που ελήφθη στους δονηστές ήταν να γίνει επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία. τις τρεις αυτές ε, επίσημα και ιδιωτικά θα επισκεφτούμε την Ταϊβάν ως προσκεκλημένη της Ταϊβάν. Ε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε δύο επίσημες επισκέψεις και για λόγους χρόνου. Και γιατί είχα την εντύπωση ότι θα μας στείλουν ιδιωτική πρόσκληση, δεν θα είναι επίσημη. Υπάρχουν προβλήματα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ε, με το ζήτημα αυτό και με το κατά πόσον ε, θα είχαμε πάρει επίσημη πρόσκληση από την Ταϊβάν λόγω ε, της τάσης ενός άλλου μεγάλου κράτους στην περιοχή. Πάντω δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, είπα και εγώ, είμαι σίγουρο ότι θα μπορούσε, ότι θα ήθελε η κυβέρνηση Ταϊβάν να μα στείλει η δυτική πρόσκληση και όσοι επιθυμούν να μπορούν να μεταβούν. Εντάξει, καλυφθήκατε. Αν δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο, για τα πρακτικά των συντονιστών. Πάντω τα έχετε μπροστά σας, κοιτάξτε τα, ε, κοιτάζετε τα κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση και πείτε μου μέχρι το τέλος. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ψηφοφορία στην έκθεση Κυρία κυρίας Τώρα, Πραγματικά η κυρία Μουσκαρδίνη έπρεπε να είναι πρόεδρο στην συνεδρίαση αλλά είπε ότι κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών και λόγω της έκθεσής της, να είμαι εγώ πρόεδρος, ε, πολύ γενναιόδορη η, πρότασή της και η προσφορά της. Πρώτα απ' όλα, έχετε όλη την κάρτα σας? Ωραία. Ξεκινάμε την πρώτη προσφορία. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά αποχές δεν περνάει. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 52 έχει υποσυρθεί. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Καταπίπτει. Μάλιστα, συγγνώμη. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία για την 57. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Όχι, το συγγνώμη. Αποχές απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Όχι, ωραία. Απορρίπτεται. 16 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ υπέρ σηκώστε τα χέρια σας κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά αυτή τη συγκεκριμένη άρχη ψηφορία Ναι, ναι, αυτό έχει ξεκαθαρίσει, ναι, τέλος πάντων. Λίγοι. Απορρίπτεται. 66. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Χωρίς... Α, unblock. Τρεις πληροφορίες unblock υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70. Χωρίς την ψηφοφορία. Σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπέρ. Εγκρίνεται. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ αποχές όχι, ζητώ συγγνώμη, λέω κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Με εκπλήτη που καταψηφίζετε, που Ντάνιελ καταψηφίζει την τροπολογία σου. Αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 και 30. Η 3 εγκρίθηκε, άρα καταπληκτή. Ωραία. 31. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Split vote on 33. First part, those... Χωριστή στην 23 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ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 37 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 αποσύρθηκε 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να το ξαναδούμε. Υπέρ. Όχι. Κατά. Απορρίφθηκε. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Δέκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έντεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δώδεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ωραία. Ψηφίζουμε την ε, πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία. Έκλεισε ψηφοφορία, έλλειψη ψηφοφορία. 3 κατά, 19 υπέρ, 2 αποχέ. Το ίδιο ε, θα κάνουμε τώρα και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματο Αρχή ψηφοφορίας. Πέρα Το ίδιο αποτέλεσμα, 19 υπέρ, 2 κατά, Δύο εποχές. Συγχαρητήρια κυρία Μουσκαρδίνη. Να συνεχίσω τις ιστορίες. Θα... Λέω πρόεδρος, θα πάρετε τη θέση μου. Oh. Yeah, yeah, I'll do all of um, this this one. Uh, This one next. Okay. Next vote is... Η επόμενη ψηφοφορία λοιπόν για την έκθεση του κυρίου Σόλτς οι εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική. Έχουμε μια συμβαστική τροπολογία, την υπαριθμό 1. Είστε έτοιμοι, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 39 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 40 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 45. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. Η 46. Υπέρ. Να το ελέγξουμε κατευθείαν ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 47 λοιπόν. Να κάνουμε το ίδιο. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Ψήφισαν όλοι. Και πάλι απορρίπτεται. Η 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη πληροφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτό. Η 50 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Έναξη ψηφοφορίας. The πέρες. Απορρίπτεται. Και άρα περνάμε στη συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 55. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Και να περάσουμε τώρα στην 61 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η παράγραφος, ε, το 62 μάλλον, τροπολογία 62 υπέρ. Κατά, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote is Πέρας. Εγκρίνεται. Η 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβιβαστική. 6. Α, συγγνώμη, η 73. Πάνω πάνω στη σελίδα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6, υπέρ. Κάτα. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 74. Κάτα πίπτη. Συμβαστική 7 υπέρ. Κάτα. Άποχες. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 12. Η 78. Και η 79. Υπέρ. Να το ελέγξουμε χρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Α, όχι, δεν ψηφίσαμε αυτή. Η 80, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 81, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμία ένσταση. Εντάξει. Να την ψηφίσουμε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 82. Καταπίπτει. Η 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 89, 90 και 92 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Να το ελέγξουμε αν θέλετε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Vote Πέρασε. Εγκρίνεται. Um, compromise. Η συμβιβαστική καταπίπτει. Και περνάμε λοιπόν στην 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 11 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 99 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Η 101 υπέρ να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote Πέρα ψηφοφορίας. Rejected. 101. 101 υπέρ. Κατά. Λέει ο πρόεδρος. Α, συγγνώμη. Να κοιτάξουμε την 102. Καταπίπτει. Και περνάμε τώρα στην συμβαστική υπαριθμών 12. Υπέρ. Καταλάβατε που ψηφίζουμε. Τη συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 108. Υπέρ. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ένα ψηφορίας. The vote Πέρας. Καταπίπτει. Η συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 117, την οποία θα τη συνδυάσουμε με τη συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 120 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α, και αποχές. Εγκρίνεται. Η 121 υπέρ. Κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2. Ενστάσεις. Υπάρχουν ενστάσεις για την προφορική τροπολογία. Να την ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 122. Υπέρ. Η 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά <laughs> Sorry. Okay, we start again. Η 124 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική υπαριθμών 3. Καμία ένσταση υπάρχει. Α, υπάρχει η ένσταση. Δεν την ψηφίζουμε λοιπόν. Η 70 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφορίας. Closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 129 υπέρ. να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 129 ενάρξη ψηφορίας. Votes closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Um, we have oral, no, uh, compromise... Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134 σε τμήματα. Στο πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote's closed. Uh, Πέρας. Απορρίπτεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 136 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140. It's split vote. First part. 140 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Υπέρ. Έναρξη ψηφοφορίας. Votes closed. Πέρες. Εγκρίνεται. Η 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 146 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. The vote's 146. για την 146. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 147. Υπέρ. Να το ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά αν θέλετε. Έναρξη ψηφορία. Πέρασε. Έγκρινεται. Η συμβαστική 17. Υπέρ. Α, συγγνώμη, ξέχασα τις δύο πάνω πάνω. Οι 149 και 151. In favor. Υπέρ. Να το ελέγξουμε. Παρακαλώ, ένα ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Compromise falls. Καταπίπτει συμβαστική και περνάμε στην 152 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 152 παρακαλώ. Έναξη ψηφοφορία. πέρασε Απορρίπτεται η 153. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά. Να το ελέγξουμε αν θέλετε. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφορίας. Closed. Πέρας. Rejected. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Η συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 18. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 22. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 25. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Compromise amendment. Η συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα. υπέρ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση που αφορά την ορολογία που χρησιμοποιείται στο ισπανικό κείμενο, έτσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω όλες ε, οι, ε, οι μεταφράσεις να ακολουθήσουν το ισπανικό κείμενο. Αναφέροντας σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς λέμε στα ισπανικά με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. In view of, εν στα αγγλικά. Αυτό δεν, δεν υπάρχει στο αγγλικό κείμενο, έτσι. Επίσης, ε, για να υπάρξει περισσότερη συνένεση, θα ήθελα να γίνει δεκτή η προφορική τροπολογία ως εξή. Να αλλάξει η έκφραση από το «good» στα αγγλικά να γίνει could. Νομίζω ότι ήταν καλύτερο να πούμε could και όχι would. Uh, uh, any Ευχαριστώ. Αντιρρήσεις, παρακαλώ. Για να γίνει το would good.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 Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε. Η πέντε Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έξι Υπέρ. Κατά. Α, καταπίπτει. Μάλιστα, συγγνώμη. Ωραία. Τώρα να ψηφίσουμε το σχέδιο της έκθεσης, ε, όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Vote Έναρξη ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τι ψηφοφορίε. Συγχαρητήρια κύριε Σούλτ. Um, Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία προς μια νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίες μπροστά σας. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Ντάνιελ, όλα εντάξει, σε βλέπω λίγο περδεμένο. Λοιπόν, συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 2, χωριστή τροπολογία σε δύο τμήματα. Με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος, μόνο το δεύτερο τμήμα, το πρώτο καταπίπτει. Ψηφίζουμε το δεύτερο μόνο τμήμα. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Ε, Δείξει παρακαλώ πολύ, σηκώστε χέρι σα καλά υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7. Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Για την 21. Άρτη ψηφοφορία. Δύο δεν έχουν ψηφίσει πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα για το σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ψηφίσατε όλοι. Δύο ακόμα πρέπει να ψηφίσουν. Ένας ακόμα. Πέρας. 23 υπέρ και μία αποχή συγχαρητήρια στον συντάκτη της γνωμοδότησης. Ολοκληρώσαμε κατά αυτόν τον τρόπο τις ψηφοφορίες και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μουσκαρντίνη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τώρα την ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ, των, ε, ε, μεταξύ τη Ευρωπαϊκή ε, Κοινότητα και των κρατών του Ειρηνικού. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτή τη συμφωνία εταιρική σχέση.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 ça simplement ah ouais. c'était pour nous un peu difficile de l'écrire. Ah oui, oui, oui, oui. Mais si vous parlez en italien, c'est... Alors, se, se gli ambasciatori, ambasciatore, il suo stato... Αν ο πρέσβης είναι έτοιμος, εντάξει, ακούτε τη μετάφραση, εντάξει. Το 2000 οι χώρες, ΑΚΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν για να ορίσουν τη νέα σχέση εμπορίας που να συμβατεί με την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου και για να τροποποιηθεί το ισχύον σύστημα των εμπορικών προτιμήσεων. Να κάνουμε λίγο όσον αφορά μια συνολική συμφωνία με την ε, ε περιοχή, ε, ελήφθη ε, μια, ε, λήφθη απόφαση για ενδιάμεση συμφωνία. Πριν από το τέλος του 2007, ε, χωρίς βεβαίως να εγκαταλειφθεί η εναλλακτική λύση για μια συνολική συμφωνία. Ε, οι δύο αυτές ε, ε, χώρες, νέα Γουινέα και Φίτζη, που είναι οι πιο σημαντικές οικονομίες, συμφώνησαν με τη συμφωνία αυτή και έχω την, την ικανοποίηση να έχουμε σήμερα κοντά μας τον Υπουργό, τον αρμόδιο Υπουργό από την Παπούα Νέα Γουινέα και τον τους δύο υπουργούς μάλλον, ε, Αλίας ε, και Εξωτερικών Υποθέσεων ε, και επίσης τον σύμβουλο στην Πρεσβεία στα Φίτζη και σας ζητώ να κάνετε μία παρουσίαση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Παππούα Νέα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά για τις σχέσεις με τα Φίτζη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας μιλήσετε για τις προσδοκίες όσον αφορά αυτή την διάμεση εταιρική σχέση και όσον αφορά τη συνολική συμφωνία. Ε, χαίρομαι λοιπόν που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας γιατί πιστεύω ότι μια ανταλλαγή απόψεων θα είναι πάρα πολύ σημαντική για τις μελλοντικέ μας σχέσεις. Το λόγο έχετε, έχει πρώτα απ' όλο ο κύριος Σαμουέλ Διαμπάλ. Uh, uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να μιλήσω εκπροσωπώντας την ε, Παπούα Νέα Γουινέα και κυρίως στον τομέα της Αλίας και έχουμε επίση μαζί μας, όπως είπατε, και τον πρέσβη της ε, περιοχής των νησιών ε, Φίτζη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να σε ευχαριστήσω καταρχάς κυρία Πρόεδρε που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε και να παρουσιάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή σας το όλο ζήτημα της ολοκλήρωσης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Ειρηνικού. Και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην τρέχουσα διαδικασία στα πλαίσια της Συμφωνίας της Λισαβόνας. Η Παππούα Νέα Γουινέα σέβεται ιδιαίτερα την ιστορική σχέση που έχει με την Ευρώπη που ξεκινάει ήδη με τους πρώτους εξερευνητές του 19ου αιώνα, καθώς επίσης και τους α, ιεραποστόλους που πήγανε στην περιοχή την δεκαετία του 50. Το 2008 άρχισε να ισχύει η Συμφωνία εταιρική σχέση, μια συμφωνία η οποία είναι δεσμευτική και προσφέρει πολύ σημαντικέ οικονομικέ ευκαιρίε στην περιοχή του Ειρηνικού, καθότι κατά αυτόν τον τρόπο πραγματοποιούνται όλε οι εμπορικέ προτιμήσει που προβλέπονται στη συμφωνία αυτή. Εναπόκειται λοιπόν τώρα στα κράτη του Ειρηνικού προκειμένου να καταφέρουν να εκμεταλλευτούν τι ευκαιρίε αυτέ που του δίνονται, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητε επενδύσει, προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικέ και οικονομικέ σχέσει σχέσεις και θεωρούμε στην Παππούα Νέα Γουινέα ότι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μπορεί να μας βοηθήσει προκειμένου να αναπτυχθούν περισσότερο τα μικρά νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού τα οποία ανήκουν στις ε, χώρες ΑΚΕ μπορεί να μην έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα από πλευράς αγοράς. παρόλα αυτά θεωρούμε ότι έχουμε καταπληκτικές πρώτες ύλε, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί μια έντονη οικονομική δραστηριότητα από την οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί όλη η κοινωνία. Μια δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην μείωση της φτώχειας, ιδίως στις πιο απομονωμένες και αποκλεισμένες περιοχές. θεωρώ ότι η εγκύτητα αυτή που έχουμε όσον αφορά τις πρώτες ύλε και η έντονη πρόσβαση που έχουμε σε αυτές δίνουν ε, μοναδικές ευκαιρίες επενδυτικές στις χώρες που θα μπορούσαν ε, να αναπτυχθούν εμπορικά, να δραστηριοποιηθούν οικονομικά στις περιοχές αυτές. Επίσης πρέπει να δερθούμε στον τομέα της ε, αλίας. Και ο τομέας αυτός αποτελεί ένα πολύ θετικό προνόμιο για την περιοχή, για όλη την περιοχή του Ειρηνικού και μας βοηθά να προωθήσουμε μια καλύτερη οικονομική περιφερειακή ολοκλήρωση. Θεωρώ ότι ο πόρος αυτός αλίας είναι πάρα πολύ σημαντικός, θα πρέπει όμως να διατηρηθεί και τις επόμενες γενιές και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται κατάλληλες πολιτικές συντήρησης των αλλιευτικών αποθεμάτων. Ακριβώς αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε την περιοχή του Ειρηνικού από την υπεραλίευση. Θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να διατηρηθούν ε, οι αλλιευτικοί πόροι προκειμένου να είμαστε σε θέση να τους εκμεταλλευτούμε και στο μέλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα μπορέσουν να αποφεληθούν ε, όλες οι πτυχές της κοινωνίας από τον τομέα αυτό και θα μπορέσουν όλοι οι νέοι αλλά και οι γυναίκες πιο συγκεκριμένα να έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας. Πρέπει να σας πω ότι ο τομέας αλίας απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες, πολύ περισσότερες από ό,τι στους πιο κλασικούς τομείς της οικονομίας. 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην Παπούα Νέα Γουινέα Πρόκειται για μια χώρα η οποία για την οποία η πρόσβαση δεν είναι πάρα πολύ ε, εύκολη, δεν υπάρχουν απαραίτητα οι ε, κατάλληλες υποδομές, η κατασκευή των υποδομών αυτών κοστίζει πολύ ακριβά. Κυρία Πρόεδρε, συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι ε, η Συμφωνία Εταιρική Σχέσης μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες και θέλουμε να αποφεληθούμε από τις από την προτιμησιακή πρόσβαση η οποία μας προσφέρεται στα πλαίσια της ε, συμφωνίας αυτής. Η παρέκκληση που προβλέπεται για τον τομέα της αλίας ε, είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση στην ε, Παππούα Νέα Γουινέα. Όπως σας είπα, το τομέα της αλίας είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Είμαστε μια νησιώτικη χώρα και χρειαζόμαστε σαφώς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, η ε, η υποστήριξή σας ήδη αντικατοπτρίζεται στις ε, εξαγωγές τόνου που κάνουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιστοιχούν περίπου στο 90% των συνολικών εξαγωγών που γίνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό είναι ένα 2%, δηλαδή οι δικές μας εξαγωγές αντιστοιχούν σε ένα 2% της συνολικής ποσότητας τόνου σε κονσέρβα που εισάγεται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι στα πλαίσια της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης θα έχουμε και στο μέλλον τη δυνατότητα να έχουμε επικοδομητικές ε, συζητήσεις και για τον τομέα της ε, αλίας αλλά και για τους υπόλοιπους τομείς της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Αυτά είναι τα πρώτα εισαγωγικά σχόλια που ήθελα να κάνω κύριε Πρόεδρε και βέβαια είμαι στη διαθεσή σα για οποιαδήποτε ερώτηση που τα μέλη τη επιτροπή σα μπορεί να έχουν ή να επιθυμούν να μου υποβάλουν. Σα ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δώσετε να πάρω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Αμπάλ και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπεν Σαμπρί. Κύριε Πρόεδρε, ήδη ο συνάδελφός μου εκφώνησε την ομιλία εξ ονόματος της χώρας μου. Δεν θέλω εγώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, αφού ακούσαμε την άποψη της ε, ε, παππού Νέας Γουινέας, θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε τον εκπρόσωπο των νησιών Φίτζη, τον πρέσβη ο οποίο έχει και το λόγο. Σα ευχαριστούμε. Thank you. Um, σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντέιβιντ Μάρτιν, ε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας να το τοποθετηθούμε για την ενδιάμεση εταιρική σχέση, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ αυτέ οι ενδιάμεσε εταιρικέ σχέσει για την περιοχή. Ε, αποτελούν αναπτυξιακό εργαλείο και ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ μα μακροπρόθεσμα. Μετά το κοτονού. Κύριε Πρόεδρε, όπω ξέρετε, η ενδιάμεση συμφωνία που, υπέγραψε το που υπέγραψαν τα Φίτζι είναι ε, μεταβατικό μέτρο έτσι ώστε να διατηρηθεί ανοιχτή η αγορά της Ευρωπαϊκή Ένωση τη εξαγωγές και να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μια συνολική περιφερειακή εταιρική σχέση. Με αυτή την έννοια η ενδιάμεση εταιρική σχέση μα έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τι ε, ε, εξαγωγέ μα ζάχαρη ε, με, με εγγυημένη ελάχιστη τιμή αναφορά μέχρι το 2012. Κύριε Πρόεδρε, να συμπληρώσω ότι παρόλο που μας εδόθη αυτή η ασφάλεια πρόσβαση στην αγορά, ακόμα δεν έχουμε αποκομίσει τα πλήρη ωφέλη της νέας ρύθμισης, διότι η παραγωγή, η ζάχαρης, αλλά και η παραγωγή, η παραγωγή της ζάχαρης, αλλά και οι εξαγωγές μας επηρεάζονται από ε, την ε, ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ζάχαρης. Μην ξεχνάτε όμως ότι εμείς ε, ως, ε, συμβα... συμβάλλον μέρος ε, του πρωτοκόλου ε, για τη ζάχαρη πρέπει να ωφεληθούμε από τα συνοδευτικά και τα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της μεταρρύθμισης στον τομέα της ζάχαρης από τον Ιούλιο του 2006 και στη συνέχεια. Η απόφαση να η, απόφαση για τη συνέχιση ε, ε, αυτής ε, της κατάστασης έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχετε κατανοήσει την κατάσταση της οικονομίας μας, δεν έχετε καταλάβει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι συνέπειες έχει στις ζωές όχι μόνο των παραγωγών αλλά και όλων όσων ζουν από την βιομηχανία της ζάχαρης και από την παραγωγή της ζάχαρης, από τον τομέα της ζάχαρης στο σύνολό της. Επίσης, ε, κοιτάξτε, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να εφοδιάσουμε ε, και, την, ε, και, το, και, το, και τη βασική μονάδα επεξεργασίας ζάχαρης στην ε, Ευρώπη. Ε, υπάρχει επίση πρόβλημα ε, που, που θα, και, και επομένω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόβλημα πρόσβαση ε, στι στις ε, ε, πρώτε ύλε. Εμεί υπογράψαμε την εταιρική, αυτή την ενδιάμεση εταιρική συμφωνία ακριβώ για να διατηρήσουμε την βιωσιμότητα του, του κλάδου παραγωγή ζάχαρη που, που είναι κρίσιμο τομέα για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών μα. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η ενδιάμεση εταιρική σχέση θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλου τομεί, όπω η Αλία, η Γεωργία και, άλλους και άλλοι τομεί τη αγορά. Για να μπορέσουμε όμω να αξιοποιήσουμε αυτέ τι δυνατότητε, απαιτούνται προσαρμογές, τεχνική συνεργασία, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι και οι μικρότερες οικονομίες στον κόσμο θα μπορέσουν να έχουν πραγματικές και ουσιαστικές εταιρικές σχέσεις με το μεγαλύτερο συνασπισμό του κόσμου, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή τα νησιά Φίτζη ε, προσπαθούν να εξασφαλίσουν το γεγονό ότι θα υπάρξουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί έτσι ώστε ε, να ακυρώσουμε και να υλοποιήσουμε την ενδιάμεση εταιρική σχέση. Αυτό σημαίνει όμω ε, ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν και οι θεσμοί και οι υποδομές έτσι ώστε να διευκολυνθεί το εμπόριο και να αξιοποιήσουμε πλήρω τι δυνατότητε συμφωνία. Τα νησιά Φίτζη εξακολουθούν να επιθυμούν ε, την, ε, τη, τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια συνολική εταιρική σχέση. Γιατί εκεί ε, συμπεριλαμβάνεται η αναπτυξιακή διάσταση που αφορά το σύνολο των χωρών ΑΚΕ στην περιοχή. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για ευάλωτες οικονομίες όπως ε, η οικονομία των νησιών Φίτζη και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, σημαντικά ε, την παγκόσμια, τις παγκόσμιες εξελίξεις και να ταχθούμε δηλαδή στην παγκόσμια οικονομία. Ελπίζουμε λοιπόν να συνεχιστεί η προσπάθεια για ενδιάμεσες εταιρικέ σχέσεις και, με και, και τελικά για μια συνολική εταιρική σχέση με όλη την περιφέρεια. Θέλουμε λοιπόν να επιληθούν τα ζητήματα τα οποία εκκρεμούν και να έχουμε ένα ισχυρό πακέτο, μια ισχυρή δέσμη μέτρων που θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια συνολική εταιρική σχέση. Οι, ε, οι, οι κανόνες καταγωγής για τα προϊόντα αλίας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα ε, γιατί η αλία είναι μεγάλη πηγή απασχόλησης ε, και βοηθά και για τη μείωση της στόχιας, κυρίως απασχόλησης γυναικών. Χαιρόμαστε γιατί αναγνωρίζεται ο μοναδικός χαρακτήρας της περιοχής του Ειρηνικού και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κίνητρο για επενδύσεις και επέκταση του εμπορίου προς το αμοιβαίο μας όφελος. Όμως τα νησιά Φίτσι δεν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις ε, διατάξεις εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν άρει ε, τους περιορισμούς τους για εξαγωγή ε, προϊόντων αλίας λόγω ορισμένων και λίγων εκκρεμών ζητημάτων στο ε, υγειονομική και φυτογειονομική φύσεω που εντόπισε ε, το Γραφείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Ε, Όμω στη συνέχεια έγιναν και άλλοι έλεγχοι και υπήρξε άρση πολλών περιορισμών στι αρχέ του μήνα. Οι αρμόδιες αρχές ε, των νήσων Φίτζη προσπαθούν να ε, ε, να χρησιμοποιήσουν ε, και να αξιοποιήσουν και, το, το συμβουλευτικό έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας στον τομέα της αλληλεία και της μεταποίηση των ελευτικών προϊόντων και ελπίζουμε να αποκατασταθεί η θέση μας ως εγκεκριμένο εξαγωγέας αλληλευτικών προϊόντων. Το, οι, την άνοιξη αυτού του έτους είπαν ότι τουλάχιστον μία εταιρεία πληρεί απόλυτε προποθέσει και θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση για έγκριση. Οι, πρόσφατες, ε, οι πρόσφατοι κτηνιατρικοί έλεγχοι ε, που έγιναν στη, ε, δεν έχουμε πάρει μάλλον το αποτέλεσμα των πρόσφατων κτηνιατρικών ελέγχων. Επίση, σα παραπέμπω στα ψηφίσματα του 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει τη μέγιστη ευελιξία όσον αφορά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για εταιρική σχέση. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της δικής σας επιτροπής να συνεχίσετε να προσέχετε ιδιαίτερα την περιοχή του Ειρηνικού, έτσι ώστε να ε, υπάρξει μια συνολική εταιρική σχέση τονίζοντα ιδιαίτερα την αναπτυξιακή σχέση που είναι ύψη τη σημασία για την περιοχή. Ένα κεφάλαιο για την ανάπτυξη που δεν αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα τη περιοχή αυτή του κόσμου δεν ωφελεί σε τίποτα. Κυρία Πρόεδρε, περιμένουμε με μεγάλη ικανοποίηση, με μεγάλη υπομονησία, συγγνώμη, περαιτέρω συζητήσει με την Επιτροπή σα, ε, καθώ θα συνεχίσονται οι διαπραγματεύσει στο άμεσο μέλλον μα ενδιαφέρει η συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσουμε την ενδιάμεση εταιρική σχέση. Διότι έχουμε περιορισμένε δυνατότητε και περιορισμένη τεχνογνωσία. Ζητούμε, σε ορισμένου τομεί λοιπόν απαιτείται συγκεκριμένη τεχνική καθοδήγηση. Καλούμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, υποστηρίξει τα νησιά ε, Φίτζη ε, και σε αυτή την προσπάθεια εγκαθίδρυσης και υλοποίησης της ενδιάμεσης εταιρικής σχέσης και ελπίζουμε να μα διευκολύνετε με μηχανισμού ε, ε, συμβούλων, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την πραγματική υλοποίηση. Τέλο, ε, κυρία Πρόεδρε, απευθύνουμε έκκληση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής σας, κυρία Πρόεδρε, να αναθεωρήσετε την πολιτική σας όσον αφορά την μη χορήγηση των επιδοτήσεων για τη ζάχαρη στα νησιά Φίτζη εάν πραγματικά ε, θέλετε όλοι, θέλουμε όλοι να εφαρμοστεί ενδιάμεση εταιρική συμφωνία, να λάβετε υπόψη ότι η πολιτική κατάσταση στα νησιά Φίτζη έχει αλλάξει ε, και ε, όπω ακριβώ άλλαξαν και οι δικές σας ευθύνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από την υπογραφή τη Συνθήκη Λισαβόνα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, σα ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μα δώσατε να κάνουμε την ομιλία αυτή και περιμένουμε με ανυπομονησία τη συνεχιζόμενη υποστήριξη. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ήταν σαφής ο λόγος σας και νομίζω τώρα ο κύριος Μάρτιν, ο εισηγητής, θα θέλει να απαντήσει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις Απευθύνομαι και στα μέλη της Επιτροπής αλλά και στους καλεσμένους μας. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο χρονοδιάγραμμα για την έκθεση αυτή. Ελπίζω να έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης στην, ε, την 9η Νοεμβρίου. Σχέδιο έκθεσης το οποίο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και θα έχουμε μέχρι τις 11 Νοεμβρίου ελπίζω τροπολογίες. Ελπίζω θα καταφέρουμε να ψηφίσουμε την 1η και 2η Δεκεμβρίου και ότι θα περάσει τελικά στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου η έκθεση αυτή. βλέπετε ότι ε, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε γρήγορα κατά αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε και ότι δεν θα κολλήσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής, ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ότι θα καταφέρουμε να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή τον Δεκέμβριο στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα αυτή τη στιγμή να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να υποβάλω και κάποιες ερωτήσεις. Εξ αρχής πάντως μπορώ να πω ότι είμαστε υπέρ της ενδιάμεσης αυτής συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Πρωτού όμω περάσω συμφωνία αυτή καθ' αυτή, θα ήθελα να Σύντομα, σε αυτά τα οποία είπε ο πρέσβης ε, των νησιών Φίτζη, εγώ όντας από την ε, άλλη πλευρά και ε, έχω έρθει σε επαφή με τους παραγωγούς ζάχαρης και κρυμμένα με την εταιρεία Tate στο, στην Αγγλία και γνωρίζω πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στα πλαίσια του τομέα αυτού και πόσο έχει πληγεί ο τομέας. Θέλω σαφώς να ληφθούν μέτρα το συντομότερο δυνατό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια, η κατάλληλη μάλλον πολιτική διευθέτηση. ό,τι έχει σημειωθεί πρόοδος, υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης και θα πρέπει κάποια συνδευτικά μέτρα να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Συμφωνούμε λοιπόν πλήρως ότι θα πρέπει τα συνδευτικά αυτά μέτρα να εγκριθούν. Το μόνο ζήτημα το οποίο απομένει αυτή τη στιγμή να, δούνε, να δούμε είναι πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή τους. Δεν τίθεται πάντως καμία αμφιβολία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, για την αγκαιότητα των μέτρων αυτών. Το, οι συνθήκες εμπορίου που έχουμε με τις ε, χώρες του ειρηνικού θα έλεγα ότι είναι αρκετά περιορισμένες ε, ουσιαστικά ένα πολύ μικρό ποσοστό του, των εμπορικών σχέσεων που έχουμε με τις χώρες ΑΚΕ αντιστοιχεί στις, ε, χώρες του Ειρηνικού, στις νησιώτικες χώρε του Ειρηνικού, στην, στο Φίτζι και στην Παππούα Νέα Γουινέα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι εμπορικές σχέσεις που έχουμε μαζί σας είναι πολύ πιο σημαντικές για σας από ότι είναι τελικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον για μας εκπροσωπούν ένα μικρό ποσοστό των συνολικών μας εξωτερικών εμπορικών σχέσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους εκπροσώπους των δύο αυτών χωρών που ήρθαν εδώ πέρα σήμερα. Μία ερώτηση που θέλω να κάνω όμω προ του καλεσμένου μα και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ακόλουθη. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέση. Σαφώ ε, ε, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα με τον τόνο και τη ζάχαρη και για την Παππούα Νεγουινέα και για τα νησιά Φίτζη. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα τα νησιά του Ειρηνικού στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρική ε, σχέση το ίμιση συγκεκριμένο το, συγκεκριμένα των νησιών επωφελείται από τη συμφωνία τα πάντα πέρα από τα όπλα και θα ήθελα να γνωρίζω από τους ε, εκπροσώπους των δύο αυτών περιοχών αν πιστεύουν ότι όντως μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης η οποία όμως να καλύπτει όλες τις χώρες της περιοχής. Ουσιαστικά να έχουμε μια συμφωνία η οποία δεν θα διχάζει την περιοχή σας αλλά θα εμπλέκει όλα τα νησιά του Ειρηνικού, όλες ε, τις νησιώτικες χώρες του Ειρηνικού. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι οι περιφερειακές σχέσεις στην περιοχή. Ήμουν εισηγητής για την Συμφωνία Οικονομικής Θερικής Σχέσης με τις χώρες της Καραϊβικής Και ένα ζήτημα το οποίο είχε προκύψει μια σημαντική ανησυχία των χωρών της Καραϊβικής ήταν ότι η υπογραφή ορισμένων χωρών μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένω να έπλητε τι συμφωνίε που έχουν με την ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν οι χώρε του Ειρηνικού φοβούνται ότι η Συμφωνία εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεάσει τι σχέσει που έχουν με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα. Επίση, ε, ένα ζήτημα που τίθεται ακόμα είναι η κοινωνία των πολιτών έχουν εκφραστεί κάποιες ε, ανησυχίες για την έλλειψη τεχνικής υποστήριξης ή ε, νομικής υποστήριξης στις προσπάθειες των χωρών αυτών να συνυπογράψουν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύουν οι χώρες αυτές ότι μπορούν ε, όντως εύκολα και ομαλά να διαπραγματευθούν συμφωνίες οικονομικής σχέσης, πολλές φορές περίπλοκες συμφωνίες οικονομικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθότι δεν ε, έχουν απαραίτητα μια τέτοια εμπειρία ή δεν εμπλέκονται σε καθημερινή βάση σε τόσο πολύπλοκες ε, συμφωνίες. Η δέκατη EDF προβλέπει υποστήριξη για προγράμματα βιώσιμης αηφόρου ανάπτυξης, αλλά θα θέλαμε επίσης να γνωρίζουμε αν η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης όντως περιέχει κάποιο κεφάλαιο το οποίο ε, θα προωθούσε περισσότερο την αναπτυξιακή συνεργασία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης προκειμένου να προωθηθούν περισσότερο τα προγράμματα οικονομικής εταιρικής σχέσης. Και επίση θα ήθελα να γνωρίζω κάτι ακόμα. Τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια του EDF ή στα πλαίσια της συνεργασίας γενικότερα προκειμένου να σας βοηθήσουμε να μειώσετε την διαρροή εγκεφάλων και δεξιοτήτων που έχετε στις δικές σας χώρες. Ξέρω και από τις συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια της κοινοβουλευτική συνέλευση ίση εκπροσώπηση Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ σημαντικές δεξιότητε και σημαντικά προσόντα για εσά που φεύγουν από την περιοχή σα. Και ένα ακόμα ζήτημα. Ε, στο παρελθόν μας επαφή με πολλούς ε, Ισπανούς ε, αλίες. Ξέρω ότι το ζήτημα της αλίας είναι πολύ σημαντικό και ξέρω και τη συμφωνία που υπάρχει για τον τόνο. Πριν από μερικά χρόνια, όταν αρχίσαμε στα πλαίσια της Επιτροπής μας να συζητούμε το ζήτημα της οικονομικής εταιρικής σχέσης, είπαμε ότι θα μπορούσε η διάταξη για την χώρα προέλευσης να γίνει λίγο πιο ελαστική. Εγώ είμαι υπέρ της εξαίρεσης που προβλέπεται όσον αφορά την ε, αλία και όσον αφορά κυρίως ε, την ε, παραγωγή, την αλία και τη μεταποίηση στον τομέα της αλίας προβλέπεται για τις χώρες του ειρηνικού Ξέρω, όπω είπε και ο εκπρόσωπο από την Παππούα Νέα Γουινέα, ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα αυτή και ότι, κατάφερε να οδηγήσει, ότι καταφέραμε κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε περισσότερε θέσει εργασία στον τομέα τη Αλία. 6.000 άτομα συγκεκριμένα κατάφεραν να βρουν εργασία στον τομέα τη κονσερβοποίηση του τόνου και μολονότι είμαι υπέρ της παρέκκλησης αυτής, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική προκειμένου να καταφέρουμε να εγγυηθούμε και την ε, αηφορία και τη βιωσιμότητα των αλλιευτικών πόρων. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο εκπρόσωπος της Παππούα Νέα Γουινέας. Μας είπε ότι ε, οι αρμόδιες εθνικές αρχές προσπαθούν να εγγυηθούν την βιωσιμότητα των αποθεμάτων τόνου στην περιοχή. Εν κατακλείδη όμως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μία διάταξη στα πλαίσια της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση υπεραλίευσης η παρέκκληση αυτή η οποία προβλέπεται αυτή τη στιγμή μπορεί και να καταργηθεί, μπορεί να αρθεί. Πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο αυτό, πάντως είναι καλό να το έχουμε κατά νου. Αυτά είχα να σας πω κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη που μακρηγόρησα. Πιστεύω ότι η Συμφωνία αυτή οικονομική εταιρική σχέση είναι πολύ σημαντική για την περιοχή του Ειρηνικού και ελπίζω θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ενδιάμεση Συμφωνία εταιρική σχέση ε, σύντομα. Το σημαντικό όμω είναι να περάσουμε από την ενδιάμεση Συμφωνία σε μια ολοκληρωμένη Συμφωνία η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επίπεδα ανάπτυξη και βιωσιμότητα για την ε, περιοχή. Και ελπίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο και δίνοντα περισσότερου πόρου, θα στεφθεί με επιτυχία το όλο Eh, Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ξεκάθαρο όλα αυτά που είπατε κύριε, κύριε Μάρτιν. Νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Αξιότιμοι κύριοι πρέσβεις. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην πτυχή της αλληλείας. Η συμφωνία σχετικά με την αλληλεία με την ε, παππούα Νέα Γουινέα ανοίγει την πρόσβαση στα προϊόντα αλληλείας της χώρας αυτής ανεξάρτητα από το τόπο όπου διεξάγονται αυτές οι αλληλευτικές ε, συμφωνίες. Αυτή η συμφωνία ασφαλώς και μπορεί να ωφελήσει την παππούα Νέα Γουινέα και την χαιρετίζω επίσης η συμφωνία αυτή πρόκειται να ρυθμίσει το θέμα της προέλευσης σε ό,τι αφορά την αλία και ε, έτσι θα προωθήσει την οικονομία της ε, Παππούας Νέας Γουινέας. Τα πλεονεκτήματα αυτά όμως θα χρησιμοποιηθούν, θα αξιοποιηθούν και από χώρες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Κίνα. Και όταν θα δοθούν αντισταθμίσεις ως προς την ε, αλληλεία και τα προϊόντα αυτά θα εισαχθούν χωρίς δασμούς ε, στην Ευρώπη, αυτό θα μας βρει αντίθετος, γιατί αυτό ασφαλώς και θα επηρεάσει αρνητικά την ε, αλληλευτική αλλά μην ξεχνάμε επίση ότι, αυτό, ότι οι κίνδυνοι θα είναι πολλοί ε, και, για την, ε, ε, και για τον κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις χώρες ΑΚΕ. γιατί υπάρχουν ορισμένε χώρες που δεν θα ωφεληθούν από αυτή τη διευκόλυνση, ενώ ταυτόχρονα κράτη-μέλη κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν πολύ σημαντική επενδυτική προσπάθεια. Σε τελευταία ανάλυση φοβάμαι ότι μόνο οι ανταγωνιστές μας θα ωφεληθούν. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα νομίζω ότι πρέπει να, να κοιτάξουμε το μέλλον. Η Παππούα και, ε, και οι υπόλοιπε ε, ε, χώρες ΑΚΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν την προμήθεια σε, αλληλευτικά προϊόντα και να επιτρέψουν τα, το, στόλο, τον αλληλευτικό στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλιεύει στην περιοχή. Η, κοινο, η κοινοτική ε, βιομηχανία πάντα τόνιζε το ενδιαφέρον της για ε, πρόσβαση στους ελευτικούς πόρους του Ειρηνικού ωκεανού. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι υπάρχουν μια, υπάρχει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και θα θέλαμε να ακούσουμε ε, από τους ε, ε προσώπους της, ε, της, της, της Παππούα Νέα Γουινέα το εξής. Πώς εξηγείται η ε, η, εξαίρεση από τους κανόνες καταγωγής όταν επιτρέπεται στους ανταγωνιστές μας να λιεύουν στην περιοχή και όχι στο στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα εγγυηθούμε την πρόσβαση του ελευτικού στόλου ε, στους σπόρους ε, του, του Ειρηνικού ωκεανού στις διαπραγματεύσεις για την εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Και τώρα, Απευθύνω ορισμένε ερωτήσει στου συναδέλφου. Ποια πολιτική πιστεύουν θα πρέπει να εφαρμόσουμε στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει εμπορικών συμφωνιών όσον αφορά την παρέκκληση από τους ε, ε, κανόνες ε, καταγωγής για τα ελευτικά προϊόντα. Και πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν, θα, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προηγούμενο ούτε να, και, και μία εξαίρεση η οποία τουλάχιστον σε μένα δημιουργεί τρομερές αμφιβολίε. Σα ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Θάλμπα. η κυρία Αντρίκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω καλώς τους ε, αξιότιμους προσκεκλημένους μας από την Παππούα Νεουίνια και τα νησιά Φίτζη. Επίσης αυτό που ανέφερε και ο εισηγητής μας, θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι η ενδιάμεση EPA αφορά μόνο ένα μικρό τμήμα του ευρωπαϊκού εμπορίου. Ωστόσο, καλωσορίζουμε την αυξημένη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εμπορικό εταίρο και θεωρούμε ότι καλύπτονται σημαντικοί τομείς όπως η πρόσβαση χωρίς τελειωνιακούς δασμούς ε, των προϊόντων από, τη, από τα νησιά Φίτζη και Παππού Νέα Γουινέα αλλά και άλλα μέτρα όπως ε, τα φυτοπροστατευτικά μέτρα. Και επίσης ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των τελωνιακών αρχών και ότι θα πρέπει ασφαλώς να υπάρχονται και ανάλογες δικλείδες ασφαλείας και για τις δύο πλευρές προκειμένου να μην υπάρχει στρέβλωση της οικονομίας. Νομίζω ότι επιθυμητό θα ήταν να καλύπτονται και άλλα θέματα που δεν περιλαμβάνονται ακόμη στις ε, τρέχουσες συμφωνίες, όπως για παράδειγμα οι διατάξεις για την ανάπτυξη, ένα κεφάλαιο για την αλληλεία, περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά θέματα, αλλά και θέματα ανταγωνισμού. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τομείς όπως ε, η φορολογία και τα πνευματικά δικαιώματα. Καλωσορίζουμε ωστόσο το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτονται ακόμα θέματα αναπτυξιακά, χορηγείται ε, από το Ταμείο Ανάπτυξη σημαντικό κονδύλιο, όπως για παράδειγμα για την βιώσιμη ανάπτυξη, για την ε, ανάπτυξη, για παράδειγμα, των οικοσυστημάτων, της βιοπικιλίας, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ο εμπορικός εταίρος θα πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε την επίτευξη του, της περιφερειακής EPA με την Ευρώπη. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξή. Για τους ειδικού κανόνες ε, προέλευσης των ε, αλληλευτικών προϊόντων. Τον έφεραν άλλωστε και οι συνάδελφοι. Έχω να απευθύνω λοιπόν κάποια ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμφωνία δεν ε, δίνει πρόσβαση στον στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα της Παππούας και των Φίτζη επειδή δεν καλύπτονται οι ανάγκες των ε, νήσων. Ρωτώ λοιπόν, τα νησιά αυτά δίνουν τέτοια πρόσβαση στην Ταϊλάνδη για παράδειγμα, στις Φιλιππίνες, στην Ταϊβάν, στην Κίνα. Η Επιτροπή έχει στοιχεία για το πώς η ενδιάμεση αυτή συμφωνία θα επηρεάσει τον ελευτικό κλάδο. Υπάρχουν ενδείξεις Πώ θα επηρεαστεί ο κλάδο κονσερβοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Τέιλορ. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω και εγώ μία σύντομη παρατήρηση σε σχέση και με το, αυτά τα οποία ακούσαμε τους συναδέλφους και τις ανησυχίες του κυρίου Θάλμπα αλλά και τις ανησυχίες πολλών ε, από εμάς σε σχέση με το γεγονός ότι η ασφάλεια ε, ε, που αισθάνεται ο καταναλωτή έχει να κάνει και με το γεγονό ότι γνωρίζει την προέλευση του προϊόντο που καταναλώνει. Άρα κάπω ε, πρέπει να συνεννοηθούν εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα νησιά Φίτζη, έτσι ώστε να καθησυχάσουμε και τον καταναλωτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που κάναν. και οι πράσινοι πρέπει να σας πω ότι σίγουρα θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω κάποιες ιδέες, φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές. Αν θα μπορούσα να σας ζητήσω περισσότερες πληροφορίες για ένα θέμα της αλληλευτικής ε, πολιτικής. Θα θέλετε να σχολιάσετε για το κατά πόσο τα οχήματα, τα σκάφη που πλέον στο είδατά σα χρησιμοποιούν όποια σημαία του ταιριάζει καλύτερα. Σημαίες ευκαιρίας. Ως ε, ευρωβουλευτή, θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο αυτό αποτελεί πρόβλημα για σας και τι μέτρα λαμβάνετε για να το καταπολεμήσετε. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι σκάφοι με σημαίε ευκαιρίας δεν αφήνουν να διευκρινιστεί η ιδιοκτησία του σκάφους. Και έτσι ο ιδιοκτήτης του σκάφους αποφεύγει τις ευθύνε του σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις συνθήκες εργασίας του πληρώματος. Και προπάντων δεν ρυθμίζεται η ελευτική δραστηριότητα του σκάφους. Κατά πόσο αποτελεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα για εσάς. ευχαριστώ και τώρα να δώσω το ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το, λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, ο κύριος Σόλτς πρώτα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τους προσκεκλημένους μας. για τη συμφωνία αυτή και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την συμφωνία αυτή και νομίζω ότι ο εισηγητής κατέστησε σαφές πόσο σημαντικές είναι αυτές οι πτυχές. σε ό,τι αφορά την ε, συνέχιση των συζητήσεων και πραγματεύσεων για μια πιο περιεκτική συμφωνία. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, αλλά να πω το εξής να αναφέρω κάτι το οποίο δεν έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο ως τώρα, αλλά ίσως και να διασαφηνίζει γιατί δεν προχωρούν οι διαπραγματεύσεις τόσο πολύ. Με τα Φίτζη, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει νόμιμη κυβέρνηση. Και αυτή η μη νόμιμη κυβέρνηση δεν μπορεί να αποτελέσει για μας εταίρο. Σε ό,τι αφορά την σύναψη δηλαδή μια αμοιβαία υποφελού ε, εμπορική συμφωνίας που θα καλύπτει κοινωνικά θέματα, περιβαλλοντικά θέματα, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακά θέματα. Και μιλάμε συχνά και μάλιστα το συζητήσαμε και χτες. Ε, συζητήσαμε για την στρατηγική του 2020 και μιλήσαμε για μια συνεκτικότητα στην πολιτική μας. Θα ήθελα λοιπόν να μας απαντήσει ο εκπρόσωπος των Φίτζη τι γίνεται με τις 103 συστάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θεωρώ προϋπόθεση για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Οι επόμενες εκλογές το 2014 Οι επόμενε εκλογέ ήταν το 2014. Αυτό θα σήμαινε για μα ότι μόνο τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, να συνεχίσουμε περαιτέρω τι διαπραγματεύσει μα και να συνάψουμε νέα σύμβαση. Αυτό δεν θα ήταν προ το συμφέρον των Φίτζη ούτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Τόμψον έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα και εγώ να μιλήσω μετά τα όσα είπαν οι εκπρόσωποι τόσο της πρεσβείας στα Φίτζη όσο και ο πρέσβης της Παππούα Νέα Γουινέας. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο προσκεκλημένους μας για την πολύ καλή ανάλυση που κάνανε της κατάστασης ανάλυση με την οποία εμείς συμφωνούμε και σας έχουμε στείλει επίσης και ένα δελτίο το οποίο κάνει μια επισκόπηση της κατάστασης στα νησιά αυτά. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε κάποια στιγμή στο παρελθόν αλλά αναφέρεται στα ζητήματα τα οποία συζητάμε, όπως για παράδειγμα η εξαίρεση για τον κανόνα της χώρας προέλευσης και υπάρχει και ένα επιπλέον τμήμα στο κείμενο αυτό το οποίο αναφέρεται στα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει στο πρόσφατο παρελθόν. Η συμφωνία αυτή αποτελεί τμήμα μιας γενικότερης διαδικασίας συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ και έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αντικατασταθούν οι διατάξεις για την προτιμησιακή πρόσβαση που προβλέπονται στα πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού και που πρόκειται να λήξουν. Και προφανώς θέλουμε να δημιουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών. Στα τέλη του 2009 όλα τα συμβαλώμενα μέρη υπέγραψαν την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ξεκινώντας με την Παππούα Νέα Γουινέα τον Δεκέμβριο του 2009. Η αίτηση όμως για τα νησιά Φίτζη ακόμα εκρεμεί γιατί προβλέπεται, μάλλον πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 76 της συμφωνίας να γίνει πρώτα μια κοινοποίηση από τα νησιά αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω αυτή τη στιγμή, κάνω μια έκκληση προς αρχές του Φίτσι, να μας αποστείλουν την κοινοποίηση αυτή το συντομότερο δυνατό. Όπως υπόθηκε η συμφωνία που έχετε ενώπιόν σας σήμερα είναι μια ενδιάμεση συμφωνία, δεν καλύπτει όλη την περιοχή και δεν περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την ανάπτυξη, ενώ περιλαμβάνει κεφάλαια που έχουν να κάνουν με, την, με υγειονομικές πτυχές, πτυχές, καθώς επίσης και διάφορα κεφάλαια που έχουν να κάνουν με την νομική φύση των πραγμάτων. Δεν θα πρέπει να θεωρείτε λοιπόν ότι πρόκειται για μια τελική συμφωνία, είναι απλώ ένα ακόμα ενδιάμεσο βήμα προς μια πιο φιλική προς την περιοχή ευρύτερη συμφωνία βασίζεται σε πρώτερες διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης και θέλουμε μέσω της συμφωνίας αυτής να προωθήσουμε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής ανάπτυξης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση επίση στην οικονομική δραστηριότητα των χωρών που θα πρέπει να ξεφύγει σιγά σιγά από την ε, απλή εξόριξη ε, πρώτων υλών. Θέλουμε επίση να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εμπορική πολιτική για την ευρύτερη περιοχή του ειρηνικού. Θα ήθελα να απαντήσω τώρα στην ερώτηση του κυρίου Μάρτιν Στόχος της ενδιάμεσης αυτής συμφωνίας είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε ε, πάυση της πρόσβασης των ε, χωρών αυτών, της προτιμησιακής πρόσβασης των χωρών αυτών στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που συμβαίνει με τις υπόλοιπες χώρες περιοχής είναι ότι είτε ανήκουν απλώς στο Everything But Arms, στο πρόγραμμα δηλαδή η πώληση των πάντων πέρα από τα όπλα, ή δεν έχουν εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα λοιπόν της ευρύτερης ολοκληρωμένης οικονομικής στερικής σχέσης της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμα στη μερίσια διάταξη, απλώς είναι ένα ζήτημα το οποίο προχωρά αρκετά αργά και πρέπει να επιληθούν πρώτα κάποια άλλα ζητήματα προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε αυτό. Πάντως σημαντική μας πρόθεση είναι όντως να έχουμε μια ευρύτερη τέτοια συμφωνία και να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε ένα κεφάλαιο αναπτυξιακή συνεργασία συμφωνία και θέλουμε επίσης και κάποια κεφάλαια που να έχουν να κάνουν και με τις ε, υπηρεσίες και με τον περιβαλλοντικό τομέα και με την ε, κοινωνική κατάσταση. Καταλαβαίνετε όμως ότι ε, σε, αναφερόμαστε τώρα σε μια περιοχή όπου η ε, οι διαθέσιμοι η δικητική ε, διοικητική δομή δεν μας επιτρέπει ακόμα να καταφέρουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα, δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε όλες τις πραγματεύσεις που θέλουμε να κάνουμε. Επίσης, πρέπει να αναφερθούμε και στις χώρες εκείνες ε, οι οποίες επιθυμούν να μπουν ε, βέβαια στην ε, συμφωνία αυτή, αλλά με τις οποίες δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εμπορική συνεργασία, δεν υπάρχει εμπόριο. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν στην ε, επόμενη φάση θα έχουμε μια βελτιωμένη εκδοχή της συμφωνίας αυτής ή αν θα έχουμε κάποιες νέες συμφωνίες. Θέλουμε επίσης να δούμε αν θα υπάρχουν νέες χώρες οι οποίες θα μπορέσουν να ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ή αν οι χώρες αυτές θα πρέπει σε μια πρώτη φάση να περάσουν και αυτές από μια ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης. Όσον αφορά τώρα για το κεφάλαιο ανάπτυξης, πρέπει να σας πω ότι ήδη γίνεται κάποια αναφορά στην υφιστάμενη συμφωνία για την αναπτυξιακή συνεργασία. Λέμε ότι θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες, προκειμένου μέσω της συμφωνίας αυτή να προωθείται και η αναπτυξιακή συνεργασία. Ένα τρίτο ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Μάρτιν είχε να κάνει με κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν ήδη οι εκπρόσωποι των ε, περιοχών αυτών. Θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων στην περιοχή αυτό, αυτή και ήδη αυτό φαίνεται στα πρώτα ανδεικτικά προγράμματα. Το ότι δεν έχουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το ζήτημα αυτό στην υφιστάμενη συμφωνία δεν σημαίνει ότι τα εθνικά και περιφερειακά αυτά προγράμματα δεν συνεχίζονται. Πρέπει να σα πω ότι τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στο IUU, δηλαδή στο πρόγραμμα αυτό που υπάρχει για την παράνομη και την ε, αδήλωτη αλλιευτική δραστηριότητα. Προβλέπεται δηλαδή και μέσω του προγράμματος αυτού μία σειρά μέτρων για την καταπολέμηση της μη βιώσιμης ή παράνομης αλίας. Και ένα ακόμα ζήτημα που θέλω να θίξω είναι ότι μολονότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή ένα ξεχωριστό κεφάλαιο όσον αφορά την πρόσβαση στις, στους πόρους, στις πρώτες αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κλάδο αυτό, σε αυτόν τον τομέα και ξέρω ότι τόσο ο Υπουργό όσο και ο Πρέσβη ε, θα έχουν περισσότερα πράγματα να πούνε για το ζήτημα αυτό. Ελπίζω ότι κατάφερα να απαντήσω στι ερωτήσει που υποβλήθηκαν. Πρέπει να σα πω επίση ότι πρόσφατα μα έφτασε μία γραπτή ερώτηση. Δεν την έχω σήμερα μαζί μου, αλλά αν δεν έχετε εσείς πρόσβαση, μπορούμε να σας δώσουμε ένα αντίγραφο της ε, απάντησής μας και αν τυχόν στην γραπτή αυτή απάντηση την έχουμε καλύψει όλα τα ζητήματα τα οποία τέθησαν σήμερα, προφανώ είμαστε στη διαθεσή για να σα δώσουμε περισσότερε διευκρινήσει. Ευχαριστώ κύριε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ιδέα λοιπόν να μα δώσετε φωτοτυπίε. Είναι προφανέ ότι τόσε πολλέ πληροφορίε δεν μπορούμε, ε, δεν τι έχουμε, δεν έχουμε πρόσβαση τόσε πολλέ πληροφορίε. Κοιτάξτε, για ε, για παράδειγμα, ε, το ίδιο πράγμα που συνέβη και με την, ε, και με την απεργία εδώ στις Βρυξέλλες. τα ανακαλύπτουμε τελευταία στιγμή. επομένως, εάν μας δίνετε έγκυρα και στις φωτοτυπίες αυτές, όλο το φάκελο μαζί και όχι έτσι κομματιαστά, εμείς θα μπορέσουμε να εργαστούμε και καλύτερα. Γιατί, κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να νομοθετήσει κανείς σε θέματα όπως ε, η παράνομη αλία. Η παράνομη αλία δεν ρυθμίζεται, δεν νομοθετείται. Απαγορεύεται και επιβάλλονται κυρώσεις. Δεν πρόκειται να τη ρυθμίσουμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μάρτιν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επανέλθω σε αυτό το στάδιο. Αλλά θα με ενδιαφέρει όμως να ακούσω κατά πόσον κάποιο από του υπουργού ή ο πρέσβης έχει να κάνει κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λοιπόν για άλλη μια φορά ε, ε, τους μας ε, και εκεί σας ρωτώ, μήπως θέλει κάποιος να ξαναπάρει το λόγο για να απαντήσει στις παρατηρήσεις που έγινε. Thank you, uh, Madam Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τα σχόλιά τους. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή David Martin για τα σχόλιά του. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους θεσμούς στο Φίτζι και νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Επιτροπής αυτής αξιότιμη κυρία Πρόεδρε μπορεί να το πράξει αυτό. Νομίζω ότι Έγινε και ένα σχόλιο για την αμοιμότητα της κυβέρνησης των Φίτζη. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει στον έλεγχό της τη χώρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα ήθελα να δηλώσω ότι η ενδιάμεση συμφωνία που υπεγράφει το 2009 υπεγράφει από την κυβέρνηση αυτή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ο αξιότιμος εισηγητής David Martin έθιξε το θέμα του τι περιλαμβάνεται στην ε, συμφωνία. Ελπίζουμε τα θέματα που δεν μας ικανοποιούν να μπορέσουν να επιληθούν στην τελική EPA. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία στην πορεία των διαπραγματεύσεων νομίζω θα μπορέσουν να ρυθμιστούν. Για θέματα ικανοτήτων, ικανότητας των Φίτζι να εφαρμόσουν τη συμφωνία, νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας, το εμπόριο και επιπρόσθετο τους πόρους. Για να βοηθήσουμε τους θεσμούς μας, την ταλωνία μας, τις αρμόδιες αρχές, για να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις των EPA για το brain drain, για την διαφυγή εγκεφάλων. Τέθηκε ένα ερώτημα. Νομίζω ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Έχουμε και εμείς αρκετούς οι οποίοι φεύγουν για τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Είναι δύσκολος ο έλεγχος των ποσοστών αυτών. Και θα είναι όλο και πιο δύσκολο στο μέλλον, αλλά θεωρώ ότι για μας είναι σημαντικό να αυξάνεται το εμπόριο αν οι βουλευτές μέσω της Επιτροπής σας, κυρία Πρόεδρε, μπορέσουν να άρουν τα εμπόδια με το εμπόριο, για το εμπόριο, είτε είναι πολιτικά τα εμπόρια αυτά, είτε οικονομικά, αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα καλυσορίζαμε. Και να επαναλάβω αυτά που είπα και άκουσα στην εισαγωγή, ότι μπορούμε να αρχίσουμε με το κεφάλαιο της ανάπτυξης. Το είπαν άλλωστε και οι αξιότιμοι βουλευτές για να ενταχθεί στην πλήρη EPA. Όπως ξέρετε, τα κονδύλια EDF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά αν ε, δεν έχουν ολοκληρωθεί προσπάθειες μέχρι το 2020, θα πρέπει να υπάρχει ένα δυνατό κεφάλαιο για την ανάπτυξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το IUU, για την παράνομη αλληλεία, θεωρώ ότι τα νησιά Φίτζη έχουν αναπτύξει την ανάλογη ικανότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει την κατάσταση. Ωστόσο δεν είμαστε ακόμα σε ιδεατό επίπεδο. Χρειαζόμαστε αρρωγή για θέματα τα οποία είναι ξένα αν θέλετε σε εμά και στις περισσότερες χώρες του ειρηνικού για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι απαιτήσει ως προς την παράνομη αλίευση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της τελικής πλήρους EPA. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα τώρα να πάρει το λόγο ο κύριος Σαμουέλ Αμπάρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τις ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου, που μου δίνετε να ξαναπάρω το λόγο αν επιτρέπετε, να ε, δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Υπουργό Αλίας, για, για ορισμένα θέματα στα οποία αναφέρθηκε. Για τις σημαίες ευκαιρίας, ευκαιρίας ε, και για, τα, για τους ελευθικούς πόρους. Ε, να δώσω το λόγο στον συνάδελφο και μετά θα μιλήσω και εγώ για τα υπόλοιπα ζητήματα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση του ε, κυρίου Θάρμα ε, για την ε, κατάσταση των αλληλευτικών αποθεμάτων. Η Παππούα Νέα Γουινέα συμβάλλει κατά 10% στην, στην παγκόσμια αλία Οι εγκαταστάσεις μας είναι ιδιαίτερα καλές και ενθαρρύνουμε ε, τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Οι εγκαταστάσεις μεταποίησης και κονσερβοποίησης είναι πάρα πολύ καλές. Όσον αφορά τώρα το κατά πόσον ο ευρωπαϊκός ε, στόλος ε, θα κατά πόσο θα μπορούσε να αλλιεύσει στην περιοχή μας, βεβαίως εμείς θέλουμε να, θέλουμε να έρχεστε, αλλά μόνο βεβαίως υπό την προπόθεση των ρυθμίσεων που ακολουθούμε εμείς στη χώρα μας. Ναι, νομίζω ότι αυτά τα δύο ερωτήματα κάνατε, έτσι δεν είναι. Μα όσον αφορά την κυρία Αντρίκενεν για τα υγειονομικά και φυτογειονομικά ζητήματα, ε, η, υπάρχει πιστοποιημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχή ε, για να εξετάζει ε, τη συμμόρφωση με τους υγειονομικούς κανόνες, ε, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην περιοχή. Σα ευχαριστούμε γιατί μα βοηθήσατε να δημιουργήσουμε αυτό το εργαστήριο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα ε, που μα βοηθήσατε. Με τη συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, φτιάξαμε τι ε, εγκαταστάσει αυτέ. Κοιτάξτε, εμά. εμείς πληρούμε τα πρότυπα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα παγκόσμια. Και αυτό θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Γιατί θέλουμε στην τελευταία ανάλυση τα ελληνικά μα προϊόντα να έρχονται στι παγκόσμιε αγορέ με, τον με σωστό τρόπο. Για να ωφελούμαστε και εμεί και να αξιούμε του πόρου μα. Να, απαντήσω τώρα αυτό το οποίο ε, ρώτησε ο κύριο Τέιλορ. για τα πλοία με σημαία ευκαιρίας. Και επίση αναφέρθηκε και στα ε, πρότυπα του, του, τη Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία. Ε, ε, να σα πω το εξή. Εμεί στην νομοθεσία μα δεν έχουμε κάτι σχετικό. δηλαδή δεν προβλέπεται κάτι για τα πλοία με σημαίε ευκαιρία. Έχουμε πλοία με σημαία δική μας που αλλιεύουν, δεν έχουμε καμία ε, ε, διάταξη για τις σημαίες ευκαιρίας. Και τώρα, όσον αφορά την απασχόληση, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες μας. 65% είναι ε, οι άνθρωποι που είναι άνεργοι στη χώρα μας. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, καταλαβαίνετε, πηγόντως. Θέλουμε να έρθουν βιομηχανίες, για να απορροφηθούν αυτές ε, οι στρατιές ανέργων που υπάρχουν ε, στους δρόμους ε, των, τόσο της πρωτεύουσας όσο και στις επαρχίες. Είμαστε μέλος του Φόρουμ του Δυτικού Ειρηνικού, στο οποίο συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμορφόμαστε και με τους κανόνες του WCFPC. Δεν ε, ενθαρρύνουμε καθόλου ε, δραστηριότητες παράνομης, αντίλωτης και λαθρέας αλίας. Ε, και μάλιστα να σας πω ότι εμείς έχουμε εγκαταστήσει ένα σύστημα παρακολούθησης σε όλα τα πλοία Κάθε πλοίο το οποίο αλλιεύει στα ύδατά μας παρακολουθείται από την αρμόδια εθνική αρχή για να εντοπίζουμε αμέσως ε, τα πλοία τα οποία ε, αλλιεύουν παράνομα. Να σας πω δηλαδή ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την ε, παράνομη αλλίευση. Επίσης. Έχουμε, έχουμε λάβει ε, έχουμε λάβει τα μέτρα έτσι ώστε να, ε, ε, να, μην, ε, να, να μην έχουμε απώλεια λευτικών πόρων από τα ύδατά μας και να μην γίνεται λαθρέα είσοδος, είσοδος λαθρέων και παράνομων πλοίων. Και μπορώ να σας πω ότι μπορείτε να έρθετε απευθεία σε επαφή με την Εθνική Αρχή Αλίας για να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μία ρύθμιση και να μπορεί να ελιεύει ο κοινοτικό στόλος, ο ευρωπαϊκό στόλος στα ύδατά μας. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δώσατε στον συνάδελφο να πάρει το λόγο, να καλύψω κανένα δύο θέματα που αναφέρθηκαν και θα ήθελα να τα επιβεβαιώσω για την απασχόληση. Η απασχόληση των γυναικών είναι πολύ σημαντική στη, στα εργοστάσια επεξεργασίας ε, ψαριών απασχολούνται κατά 80% γυναίκες οι οποίες ε, προέρχονται από, τις, ε, από την Ήπεθρο λόγω οικονομικών προβλημάτων και είναι σημαντικά τα χέρια αυτά γιατί δεν έχουν πολλά δεν υπάρχουν πολλές άλλες θέσεις εργασίας σε, άλλες, σε άλλους κλάδους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν, καθώς και η προετοιμασία ε, των ψαριών για κονσορβοποίηση. Απασχολούνται πολλές γυναίκες εκεί. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο απάντησε και ο συνάδελφος για την δυνατότητα των ευρωπαϊκών στόλων να αλλιεύουν στα ύδατά μας. Καλωσορίζουμε τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στα πλαίσια του PNG. Uh, uh, Στην Παππούα Νέα Γουινέα καλωσορίζουμε τις ευρωπαϊκές επενδύσεις Θα θέλαμε έτσι να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και θεωρώ ότι επειδή οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΚΕ έχουν ιστορία 30 και πλέον χρόνων, αυτό μας δίνει πολλές ευκαιρίες. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τη νέα συμφωνία, η οποία θα είναι περιεκτική. Με τις ρυθμίσεις αυτές, στο μέλλον θα καλωσορίσουμε το στόλο σας μαζί με τις επενδύσεις σας και τη τεχνογνωσία σας. Δεν θεωρώ ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα. Καλώς να ορίσει ο Ευρωπαϊκός Στόλος και οι ευρωπαϊκές επενδύσεις. Για τους ε, κανόνες προέλευσης, Αυτό καλύπτεται στις ε, σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΜΟΝ. Σε ό,τι αφορά τώρα το γεγονός ότι συμφωνούμε να συμπεριληφθούν και αναπτυξιακές ε, πτυχές στην ε, συνεργασία, όπως και τα, οι πτυχές που αφορούν το περιβάλλον, την πνευματική ιδιοκτησία κτλ. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα Ένα από τα προβλήματα για τη σύναψη συμφωνίας ήταν ότι πολλές νησιωτικές χώρες πολλές φορές δεν είναι σε θέση να καταλάβουν απόλυτα το τι συμβαίνει και να το ελέγξουν. Όπως είπατε, θα θυμάσαστε κυρία Πρόεδρε, το 2008 η χρονική συγκυρία των διαπραγματεύσεων ήταν πάρα πολύ σημαντική και τα νησιά Φίτζη δραστηριοποιήθηκαν έντονα. επιβεβαιώθηκε τότε η σωστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χαρήκαμε που συνέχισαν οι διαπραγματεύσεις. Θα ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή που βοήθησε προς την κατεύθυνση αυτή. Συμφωνούμε ότι η συνεκτική EPA θα ήταν πολύ καλύτερη για να τεθεί σε καλύτερη βάση η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προωθηθεί και η περιφερειακή συνεργασία. Έχουμε συζητήσει και με άλλες νησιωτικές χώρες, τις έχουμε ενθαρρύνει να υπογράψουν, αλλά σε γενικέ γραμμέ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι για πολλέ νησιωτικέ χώρε δεν υπάρχει ουσιαστικά εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα Φίτζη υπάρχει σχέση προς την αλληλεία και τη ζάχαρη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική επιβίωσή μας. Γι' αυτό λοιπόν και προσυπογράψαμε και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κατανοήσει τη σημασία των συμφωνιών αυτών. Η αλληλεία μπορεί να αντιστοιχεί στο 2% της ε, αγοράς σας, αλλά για την Παππούα Νέα Γουινέα αντιπροσωπεύει 95% της συνολικής μας αγοράς των εξαγωγών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, όπως και γενικότερα η απασχόληση. Άρα, στο σημείο αυτό, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι επιβεβαιώνουμε ότι πρόκειται για σημαντικό οικονομικό ζήτημα για τη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Και ελπίζουμε ότι οι αξιότιμοι βουλευτές όταν θα εξετάσουν το θέμα αυτό το Δεκέμβριο θα συνειδητοποιήσουν και θα αντιληφθούν την οικονομική σημασία του θέματος αυτού για την Παππούα Νέα Γουινέα και για τις υπόλοιπες νησιωτικές χώρες για τον τόνο αλλά και για τα υπόλοιπα αλληλευτικά προϊόντα και θα ελπίζουμε ότι θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πρόσβαση στην αλία. Ακόμα και αν είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε προσυπογράψει για την ε, εξαίρεση αυτή. Ήταν επειδή εμείς ξεχωρίσαμε τότε που δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών του Ειρηνικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταλάβετε, ελπίζω, πόσο σημαντικό είναι το μέσο αυτό για τις οικονομίες μας. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε τους υπουργούς και την εξοχότητα ε, του τον πρέσβη. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Σόλτς για να μιλήσει για λίγο. Σας υπενθυμίζω πρέπει να είστε πάρα πολύ σύντομος γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος κυρία Πρόεδρε. Φαντάζομαι πάντως ότι το ζήτημα το οποίο συζητάμε είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και είναι σημαντικό τουλάχιστον υπάρχει μια κοινή προσέγγιση και θα ήθελα απλώς να τονίσω την απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπος των νησιών Φίτζη Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι βρισκόμαστε στην μετά Λισαβόνα εποχή και σε σχέση με το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραματίζει πλέον ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εμπορικών συναλλαγών και των εμπορικών σχέσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι εμείς προφανώς θέλουμε να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατανόηση της κατάστασης στη χώρα σας και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε με την Συμφωνία εταιρική Σχέσης. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και θα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση και μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον κύριο Βέλντερ που δεν είναι εδώ. Ε, Μικρή σύγχυση που σημαίνει και αυτό κάποια φορά. Ε, να μιλήσετε για το επόμενο θέμα. Οπότε τελειώσαμε εδώ ε, με τις ε, παρεμβάσεις. Σας θυμίζω το χρονοδιάγραμμα πριν από τις 9 Νοεμβρίου για ε, ανταλλαγή απόψεων εκ νέου ε, πάνω στην έκθεση αυτή 11 Νοεμβρίου τροπολογίες ψήφο στην Επιτροπή 2 ε, Δεκεμβρίου και ολομέλεια του, το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Θα δούμε, ανάλογα με το πώς θα πάμε το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε τους προσκεκλημένους μας και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η τροποποίηση του κανονισμού 732 του 2008 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικών δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2011. Η κοινότητα ε, παρέχει αυτές τις ε, ε, προτιμήσεις στα πλαίσια των γενικευμένων προτιμήσεων. Από το 1971 σας υπενθυμίζω. Πρόκειται για μια εμπορική ρύθμιση που ακολουθεί αυτό το οποίο ήδη είχε δώσει ε, η κοινότητα ε, σε 176 χώρες αναπτυσσόμενες υπό τη μορφή μειωμένων ε, δασμών. Ο κανονισμός γενικευμένων προτιμήσεων αυτή τη στιγμή θα εκπνεύσει την 31η Δεκεμβρίου του 2011 το 2008 που ενέκρινε το ισχύον σύστημα είχε δώσει εντολή το Κοινοβούλιο να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για την περίοδο που θα ακολουθήσει τον Ιούνιο 2010. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμα υποβάλει προτάσεις αναθεώρησης, αλλά πρόταση παράτασης ε, του υφιστάμενου κανονισμού μετά την 21η Δεκεμβρίου 2011. Αφού ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση το Μάρτιο, η Επιτροπή προέβλεψε να υποβάλει την πρόταση ε, για την αναθεώρηση του κανονισμού μετά το 2011, ε, δηλαδή τότε να υποβάλει την πρόταση και στο μεταξύ ε, να, να, να ισχύει ο φυστάμενο κανονισμό και να υπάρχει απαραίτητο χρόνο στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για να συμφωνήσουν ε, σε μια νέα ρύθμιση που θα ακολουθήσει την ε, συνηθισμένη ε, νομοθετική διαδικασία. Αυτό είναι ο λόγο που για να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια του, του ισχύου του συστήματο παρουσίασε ένα κανονισμό για ανανέωση, για παράταση, για να μην υπάρξει νομική αβεβαιότητα. αβεβαιότητα. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Σόλτ, να μας εξηγήσει το ζήτημα. Σας δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, συνάδελφοι, αγαπητοί πρόεδρε, αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώς όλοι γνώριζετε καλύτερα τους μηχανισμούς GSP+, από ότι εγώ, γιατί εγώ δουλεύω ως Ευρωβουλευτής ε, μόλις ένα έτος. Αλλά να σας επιστήσω την προσοχή στο πώς γεννήθηκε, πώς προέκυψε το εργαλείο αυτό. Να σας δώσω κάποιες πληροφορίες ε, που θα μας βοηθήσουν να κοιτάξουμε τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Μιλάμε για γενικευμένες προτιμήσεις. Πρόκειται για ένα κλασικό εργαλείο προς τις αναπτυσσόμενες χώρες δηλαδή να μην υπόκεινται στους συνηθισμένους δασμούς οι αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό έχει μακρά ιστορία ως εργαλείο. Το 1968 έγινε σύσταση για τη δημιουργία ενός συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων προς τις ανυπτυσσόμενες χώρες από τις ε, εκβιομηχανισμένες χώρες σε μη αμοιβαία βάση. Έκτοτε οι χώρες του ΩΣΑ έχουν εφαρμόσει τέτοια συστήματα μη αμοιβαιότητας, μη αμοιβαίας ε, σχέσεις, αλλά και διμερεί, διμερείς αμοιβαίες συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφήρμοσε το 1971 για πρώτη φορά τέτοια συστήματα. Τρεις τύποι τέτοιες, ε, τρεις τύποι τέτοιας ε, βοήθειας υπάρχουν. Καταρχάς, όταν ε, απολαμβάνουν όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες τέτοια ωφέλη. Κατά δεύτερον, το GSP Plus που προβλέπει επιπρόσθετα ωφέλη για χώρες που πληρούν κάποια διεθνή πρότυπα. Και αυτό περιλαμβάνει μια συνεκτική πολιτική. Μιλάμε κυρίως για εργασιακά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, καλή διακυβέρνηση, περιβαλλοντικά πρότυπα και το καθεξής. Και τρίτη, τρίτος τύπος είναι η πρωτοβουλία όλα εκτός από όπλα για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Άρα γενικά το σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν οι πιο πολλές αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν μας ε, βοηθάει να καταλάβουμε με το, το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. το 2001 αναπέμφθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας της ε, διαβούλευσης το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο. Οι βασικές διατάξεις του GSP δεν άλλαξαν, αλλά σκοπό είχαν να διευκολύνουν την εφαρμογή του συστήματος. Στις 21 του Δεκεμβρίου του 2007 παρουσιάστηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2008 31 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο να δώσει την γνωμοδότησή του μέχρι το 2009. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο δεν είχε το χρόνο τον απαραίτητο να καταρτήσει γνωμοδότηση και πρόκειται για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ήταν πάρα πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα τότε. Στο ψήφισμα της 5ης Ιουνίου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ρητά ότι δεν είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι στο μέλλον θα πρέπει να έχει πιο πολύ χρόνο το Κοινοβούλιο για να διαδραματίσει σωστά το ρόλο του και αναφέρεται ή αναφέρει το ψήφισμα ότι η πρόταση ε, αναθεωρημένου ψηφίσματος από το Ιανουάριο του 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 θα την δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι 1η Ιουνίου 2010. Αυτό τι σημαίνει ότι το τρέχον ε, σύστημα θα εκπνεύσει 31 Δεκεμβρίου του 2011 και αυτό σημαίνει ότι στις 26 Μαΐου η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε την πρόταση που εξετάζουμε. Ωστόσο, η πρόταση αυτή περιλαμβάνει νέου κανονισμού θα αποτελέσει ουσιαστικά μία παράταση του υφιστάμενου κανονισμού. Και συγχωρέστε με για το μακρύ αυτό ιστορικό, αλλά στο ψήφισμα του 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να γίνει μελέτη αντικτύπου για τις επιπτώσεις του GSP από 1η Ιανουαρίου του 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 και αυτό μέχρι το Μάρτιο του 2010. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω το υλικό αυτό. Δεν ξέρω αν έχει διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο αυτή η μελέτη που Ο τρέχον κανονισμός ε, παραμένει απαράλλαχτος. Ο κανονισμός ο οποίος είχε τεθεί σε εφαρμογή για τρία χρόνια και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αντικτύπου προτού καταρτιστεί ο νέος κανονισμός. Εν ώψη της προετοιμασίας νέας πρότασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010 ε, κύκλο νέων διαβουλεύσεων. Θα πρέπει να συλλεχθούν στατιστικά στοιχεία, να γίνουν μελέτες αντικτύπου. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υπόλοιπη περίοδος για την εφαρμογή του κανονισμού GSP είναι υπερβολικά σύντομη προκειμένου να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια νέα πρόταση για νέο κανονισμό και να μπορέσει να συμφωνήσει και το Κοινοβούλιο με την ε, σωστή νομοθετική διαδικασία πριν το τέλος του 2011 και γι' αυτό έγινε πρόταση να παραμείνει ως έχει κανονισμός, να γίνει rollover. Το οποίο τι θα σήμερα με τη σειρά του, ότι η κατάσταση θα έπρεπε να πάρει παράταση για δύο χρόνια. Ωστόσο, και τώρα περνάω στην πραγματική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας έχουν ε, ενισχυθεί οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και έχει πλέον λόγο το Κοινοβούλιο για την ομιμότητα, τον κατάλογο των ε, χωρών, των χωρών που υποφελούνται από το GSP σε ό,τι αφορά τον προσωρινό ρόλο των ε, ρυθμίσεων κτλ. Αν λοιπόν ο τρέχον κανονισμό εκπνεύσει το 2011, δύο χρόνια μετά τη θέση σε λειτουργία τη εφαρμογή της συνθήκη τη Λισαβόνα, με την προτινόμενη παράταση η κατάσταση θα πάρει άλλα δύο χρόνια παράταση. Τουλάχιστον μέχρι τέλη 2013, τέσσερα χρόνια δηλαδή μετά από τη θέση σε εφαρμογή, σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και να σας πω με πάσα ειλικρίνεια ότι δεν θεωρώ ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να αποδεχτούμε την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προτείνω τροπολογίες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διασφαλίσουμε ότι οι νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Λισαβόνα θα ληφθούν υπόψη μετά το 2011. Ένα άλλο σημαντικό θέμα consider the Pakistan Ένα άλλο σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι πίεση ασκείται από την πραγματική κατάσταση. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος στις χώρες αυτές. Και φυσικά μας το έθεσαν αυτό το θέμα και το Συμβούλιο να επιτρέψουμε και στο Πακιστάν να ωφεληθεί από το GSP+. Σε αυτό έχουν συμφωνήσει τα κρατημέλη σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές από το Πακιστάν για να ε, βοηθηθεί η οικονομική ανάκαμψη της χώρας εκ παραλίλου. Το GSP δέχεται τα πειρά της κριτικής και από τις χώρες που ωφελούνται από το GSP και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, γιατί πολύ συχνά εξαιρούνται τμήματα των χωρών από τις πιο επωφελείς διατάξεις. Χώρες οι οποίες ε, μπορεί να ωφεληθούν από τις προτιμήσεις δεν είναι αυτέ οι οποίε απαραίτητα σύμφωνα με του όρου του GSP θα έπρεπε να αφαιρεθούν. Και πάλι αυτό το παράδειγμα του Πακιστάν. Φυσικά όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και μία δυνατότητα που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δώσει στο Πακιστάν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, το οποίο θα ήταν μία μικρή διόρθωση της νομιμότητας, των κριτηρίων νομιμότητας του GSP. Σήμερα οι χώρες δεν μπορούν να ωφεληθούν από το GSP αν εκπροσωπούν ποσοστό άνω του 1% της ευρωπαϊκής ε, αγοράς. Το Πακιστάν υπερβαίνει σαφώς το ποσοστό αυτό. Άρα, αν το 1% γίνει 1,5%, 2% μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Αυτό θα έδινε στο Πακιστάν πολύ καλύτερη πρόσβαση στην αγορά. Και θα ήθελα να μου να ακούσω τις ε, γνώμες της υπόλοιπης Επιτροπής, να ακούσουμε και τους συντονιστές μας. Εν ώψη και όσων υπόχθηκαν και συζητήθηκαν την Άνοιξη του 2010, για να μην μακρηγορήσω, κυρία Πρόεδρε, να πω το εξής. Να θέσω κάποια ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και προς τους συναδέλφους. Πότε θα έχουμε στα χέρια μας την έκθεση αντικτύπου. Πότε θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβόλευση. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ε, υποβάλει τις θέσεις τους. Θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει τα ανάλογα στοιχεία. Ένα άλλο ερώτημα. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο σχεδίασε μία έκθεση η οποία τελικά εγκρίθηκε και έγινε ο τρέχον κανονισμός. Δεν είχαν λεφθεί τότε πολλά από τα σχόλια του Κοινοβουλίου. Γιατί μπορεί να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τρίτον, ξέρουμε ότι η μεταρρύθμιση του GSP είναι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πότε θα ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των κανόνων προορισμ, ε, καταγωγής. αναφορικά με τα GSP. Και, τρίτο, και τέλος, θα ήθελα ως Επιτροπή να ζητήσουμε από την νομική υπηρεσία να μας πει αν θα μπορούσε να γνωμοδοτήσει για τις αλλαγές στον κανονισμό του GSP για τις αλλαγές που χρειάζονται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αυξημένη αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου όπως ορίζεται από τη ε, Συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ και ε, εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να τηρήσουν το χρόνο που έχουν διαθεστεί τους. Διαφορετικά δεν θα προλάβουμε, δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι κύριος Κάτφελερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν ε, ολοκληρώσε το έργο της έγκαιρα και ακριβώς για αυτό το λόγο Τώρα μιλάμε για την παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος. Θα ήταν καλό να μας πείτε γιατί δεν μπορέσατε να προετοιμάσετε ένα νέο σχέδιο έγκυρα. Ποιοι είναι οι λόγοι για αυτή την καθυστέρηση. Τώρα αυτής της κατάστασης δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να δεχθούμε το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τη νέα πρόταση όσο να πιο γρήγορα γιατί πιστεύω ότι ο κανονισμός αυτός ε, περιέχει ε, κάποιες αντιφάσεις και οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν συγκεκριμένα ερωτηματικά. Για παράδειγμα, γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που ίσως είναι οι πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο. Γιατί να τους ενισχύουμε ενώ άλλες χώρες, πολύ πιο φτωχές, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τέτοιες εμπορικές δυνατότητες. Άλλη ε, ε ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών. Σε σχέση με τις ε, χώρες BRIC, ε, ε, Βραζιλία κτλ. παίρνουν ε, ενώ παίρνουν χρηματοδότηση, από την άλλη παραβιάζουν συμφωνίε. Η Κίνα ε, είναι ο μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο και ε, με νομισματικά κόλπα δημιουργεί κίνδυνο σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Και υπάρχουν και προβλήματα με τι εξαγωγέ των χωρών που εμεί θέλουμε να υποστηρίξουμε το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων. Γι' αυτό σα παρακαλώ, σκεφτείτε τα συμφέροντα των φτωχότερων χωρών και προχωρήστε έγκαιρα στην αναθεώρηση. Βρείτε τρόπου για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ένα νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, με ένα μεταρρυθμισμένο σύστημα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. David Martin έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Βίτο Μερένιο και ο δισηγητή από του σοσιαλιστέ δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μα. Μου ζήτησε πάντω εξ ονοματό να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Θα είμαι σύντομο καταρχάς συμφωνεί και με άλλους και λέει ότι λυπάται που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να υποβάλει εγκαίρως μία πρόταση για ένα νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων προκειμένου το νέο αυτό σύστημα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν τήρησε δηλαδή το χρονοδιάγραμμα το οποίο έπρεπε να έχει προβλεφθεί και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2010. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν να υποβάλει μια νέα πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναθεωρήσουμε εξ ολοκλήρου το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Το νέο σύστημα θα πρέπει να απευθύνεται περισσότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η μη τήρηση του χρονοδιάγραμματος αυτού είχε αρνητικές επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και προσπαθούμε με τη βοήθεια του εισηγητή να καταλήξουμε τελικά σε μία συμφωνία για την παράταση του ε, υφιστάμενου κανονισμού. Θα πρέπει πάντως ο κανονισμός, ο νέος, να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατό. Αυτά ήθελα να πω ε, εξ ονόματος του Σκιώδου Σιγητού από τους Αλιστές. Για το Πακιστάν τώρα εγώ ίδιος θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε τη χώρα αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια περιεκτική πλήρης αναθεώρηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μια νέα συμφωνία για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και αυτή να ισχύει στην περίπτωση του Πακιστάν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μπέρνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να υπάρξει ρόλο αυτό και η παράδαση του κανονισμού. Φυσικά αυτό θα πρέπει να γίνει με τον πλέον σωστό και κατάλληλο τρόπο. Γιατί αν μας πάρει πάρα πολύ χρόνο στο Κοινοβούλιο και παρατείνουμε υπερβολικά την ε, κατάσταση, ο κίνδυνος είναι τελικά να μην έχουμε από 1η Ιανουαρίου 2012 νέο κανονισμό και να υπάρχουν νέα εμπόδια βασμολογικά για τις φτωχές χώρες. Και νομίζω ότι να προσέξουμε να μην υπάρχει ε, αγώνας για, μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για το ποιο θα επικρατήσει. Μου προκαλεί κάποια νευρικότητα αυτά που μας ανέφερε ο εισηγητής, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία να επιδείξουμε ότι πρόκειται ότι είμαστε ένα όργανο το οποίο λαμβάνει σοβαρά τις ευθύνες του σε ό,τι αφορά τις τιμές κατόφλι τώρα που ανέφερε και ο εισηγητή για την ε, συμμετοχή στο GSP+. Αυτό το συζητήσαμε τη μακρόν. Κατά πόσο το 1% είναι η σωστή τιμή ή όχι. Ακούσαμε πολλές και διαφορετικές γνώμες και νομίζω ότι ήταν πολύ ε, οριακό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Συμβούλιο των Υπουργών. Νομίζω ότι Υπάρχουν λόγοι για να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό και αυτό δεν εξαρτάται νομίζω μόνο από το Πακιστάν. Χρειάζεται ούτως ή άλλως αυτή η αύξηση. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το Πακιστάν επηρεάζεται σαφέστατα γιατί βρίσκεται στο 1,2% και όχι στο 1%. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια καλή ευκαιρία για μας να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται για να αλλάξουμε την τιμή αυτή, το ποσοστό αυτό. Και πού θα γίνει, πότε θα το κάνουμε αυτό, αν όχι τώρα. Τι άλλα εμπορικά εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αν θέλουμε να περιμένουμε έως το 2014 για να αλλάξουμε αυτές τις ε, τιμές, θεωρώ ότι θα χάσουμε μια χρυσή ευκαιρία να διευκολύνουμε κάπως το Πακιστάν. Αν λοιπόν ξέρουμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε αυτή την τιμή κατόφλη, γιατί να περιμένουμε, γιατί να χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Ωστόσο, θα πρέπει να επιδείξουμε προσοχή, να μην αλλάξουμε υπερβολικά πολλά στοιχεία και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός τελικά θα προκύψει το συντομότερο δυνατόν προκειμένου οι ιστορικέ μα διαδικασίε να μην επηρεάσουν τι φτωχέ χώρε. Ευχαριστώ. Ο κ. Κάσπαρη έχει το λόγο αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Σόλτς για την πολύ καλή εισαγωγή που έκανε στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι μας βοήθησε ιδιαίτερα αυτό. Βλέπουμε ότι συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Στο Κοινοβούλιο ψηφίσαμε το αντίστοιχο ψήφισμα και νομίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο έχουμε απέναντι μας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γκλάτφελντερ και οι υπόλοιποι μίλησαν για τη σημασία του νέου κανονισμού. Για κάποια θέματα συμφωνώ. Για παράδειγμα, αυτά που είπατε για τα κράτη του Περσικού κόλπου με βρίσκουν σύμφωνο. για πολλά θέματα δεν χρειάζεται περαιτέρω διαπραγματεύσεις γιατί ρυθμίζονται ούτως ή άλλως από το GSP. Ωστόσο αυτό δεν είναι συμπεριφορά εμπορικών εταίρων και ε, ίσως λοιπόν θα έπρεπε όντως να έχουμε πιο σκληρή στάση έναντι κάποιων εμπορικών εταίρων και να τροποποιήσουμε τις GSP αλλά αφετέρου θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ γρήγορα πού βρισκόμαστε σήμερα. Βρισκόμαστε τον Οκτώβριο του 2010 και αυτό τι σημαίνει ότι όσο του καταλήξουμε σε μία νέα ρύθμιση η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή έχουμε 15 μήνες μπροστά μου και μιλώντας και με τους εκπροσώπους των χωρών που εμπλέκονται και μιλώντας με τους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού κλάδου μιλάμε για συμβάσεις μισού έως ένα έτους. Τέτοιες συμβάσεις συνάπτουν οι φορείς αυτοί. Είναι σημαντικό λοιπόν για όλους να ξέρουν τι μπορούν να υπολογίζουν, τι θα δεθεί σε εφαρμογή από το 2012, γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο αν κάποιες ε, εταιρείε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναγκαστούν να καταγγείλουν συμβάσεις που έχουν συνάψει. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ ατυχής η συγκυρία, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα παραταθεί η ο υφιστάμενος κανονισμός και να μην κάνουμε αυτό που πρότεινε εν μέρει ο εισηγητής, να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες για να τις τροποποιήσουμε. Θα πρέπει το χρόνο που έχουμε μπροστά μας να τον αξιοποιήσουμε όταν θα έχουμε και τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου και της ε, διαβούλευσης, να κάτσουμε και να δούμε πώς τα προβλήματα τα οποία εντόπισαν οι συνάδελφοι μπορούν να επιληθούν από 1η Ιανουαρίου 2014 θα πρέπει να υπάρχει νέα, νέος κανονισμός. Και πέρα από τη συνθήκη της Λισαβόνας, κύριε Σούλτς, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε χρόνο για να κοιτάξουμε την ποιότητα της νομοθεσίας, την αξιοπιστία των συστημάτων αυτών. Όλα αυτά είναι σαφώς πιο σημαντικά και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε ανάγκη, που χρειαζόμαστε κατά το 2011. Αν τα καταφέρουμε το 2011, μπορεί να προκύψει ο νέος ε, κανονισμός το 2012, γιατί και όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν 1,5 χρόνο στη διάθεσή τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους τους φορείς, αλλά και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ευχαριστώ κύριε Κασπάρη. Και επιτρέψτε μου να συμφωνήσω με την ανάλυση σας. Κύριε Στέρντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα σας δημιουργεί έκπληξη ότι συμφωνώ και με τους τρεις ε, εκπροσώπους του ΕΛΚ. Ντέιβιτ, με ανησυχεί κάπως η θέση για το Πακιστάν. Για μένα, το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων έχει ως στόχο να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και το Πακιστάν ε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι υπάρχουν ευκαιρίες πραγματικά ε, έτσι ώστε το, το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων, το ενισχυμένο, ε, θα τους βοηθήσει. Ε, βεβαίως υπάρχει μια κατάσταση ε, κρίσιμη και πρέπει... Ναι, ναι, ναι, πάρε το λόγο. Όχι, να ξεκαθαρίσω. Ότι θα προβούμε σε αναθεώρηση του GSP+, ε, ελπίζω το Πακιστάν να αποτελέσει μέρος της νέας συμφωνίας. Εγώ μιλώ για την προσωρινή συμφωνία και ρυθμίση για μια χώρα. Θα υπάρξουν άλλα προσωρινά μέτρα που θα βοηθήσουν το Πακιστάν. Δεν λέμε να αποκλειστεί και από το καινούριο σύστημα, αλλά να περιμένουμε ε, το 2012. Μάλιστα. Ωραία. Να τελειώσει ο διάλογο. Κοιτάξτε. Κύριε Σούλτ, εσεί βάλετε το Πακιστάν συζήτηση. Πρώτα συμφωνώ με τον Κρίστοφερ και με τον Ντάνιελ. θα πρέπει εδώ να δούμε ε, το κατόφλι. Γιατί η συνολική αρχή του GSP Plus είναι να βοηθήσει ε, τις χώρες αυτές και να δώσουμε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει ότι βοηθά τις αναψώμενες χώρες έτσι ώστε να ωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες. Επίσης, και εδώ ίσως αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ανησυχώ ιδιαίτερα για το γεγονός ότι αφαιρέσαμε τη Σρι από το σύστημα. Καταλαβαίνω του λόγου του οποίου έγινε αυτό, αλλά και εδώ έχουμε μια χώρα η οποία ε, αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια. Εμφύλιο πόλεμο που ήταν καταστροφικός για τη χώρα και επειδή εγώ έχω δει και στη δική μου χώρα εμφύλιο πόλεμο ε, με τον Ήρα κοιτάξτε τελικά καταφέραμε να βρούμε μια λύση οπότε ε, και εδώ στη Σρι θα υπάρξει λύση. Γι' αυτό ελπίζω να, τα ξα... ξανασκεφτεί το ζήτημα η Επιτροπή. Ε, είμαι απογοητευμένο λοιπόν που δεν έχει δώσει απάντηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ξαναλέω, εδώ έχουμε μια ευκαιρία να βοηθήσουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυσσόμενε χώρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στέρντι. Βεβαίω. Νομίζω ότι εξετάζοντα το πρόβλημα αυτό πρέπει να ξαναγυρίσουμε και να αρχίσουμε να εξετάζουμε τι έχει συμβεί και στην περίπτωση τη Σρι Ο κύριος Αρίφ έχει το λόγο. Νομίζω ότι ε, ο Ντέιβιντ είπε ποια θα μπορούσε να τα γενικότερα η στάση μας, η στάση της ομάδας μας στο GSP. Όσον αφορά τώρα το Πακιστάν, καταλαβαίνω ότι λέει ο κύριος Στάρντι για το GSP+, ότι θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιες χώρες το σύστημα αυτό προκειμένου να πτυχθούν. Ωστόσο το GSP Plus προσφέρεται έναντι κάποιων δεσμεύσεων των χωρών αυτών που θα πρέπει να τηρούν κάποιες σημαντικές συμβάσεις σε διεθνές επίπεδο. Συμβάσεις που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα συγκεκριμένα και δεν μπορούμε εμείς με την επίφαση ότι βοηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο τις αναπτυσσόμενες χώρες να ξεχνάμε τις βασικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μας και δι' τις εμπορικές μας σχέσεις. Συμφωνώ λοιπόν ότι μπορούμε όντως να προβλέψουμε συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουμε το Πακιστάν. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να προβλέψουμε εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις ακόμα και στα πλαίσια του ΠΟΕ, αλλά το να ανοίξουμε εντελώ τη συζήτηση και να πούμε ότι καταρρύπτουμε όλες τις προποθέσεις που έχουμε θέσει για τις υπόλοιπες χώρες για να βοηθήσουμε το Πακιστάν, τότε ξεχνάμε ουσιαστικά αυτά τα οποία θέτουμε ως προποθέσει στα πλαίσια του GSP. Θα ήμουν λοιπόν ο ίδιο ιδιαίτερα προσεκτικό. Κοιτάξτε, ναι, όταν θα έχουμε ένα νέο κανονισμό μπορούμε το ζήτημα αυτό να το θέσουμε εκ νέου. Πιστεύω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινήθηκε καλά απέναντι στη Σρι Λάνκα, να απόκειται στην κυβέρνηση της χώρας αυτής να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα και να δώσει κάποιες ε, εγγυήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταφέρει να αποφεληθεί εκ νέου από το GSP. Και μόνο ότι διαφωνούμε πολλέ φορέ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έλεγα εγώ ότι αυτή τη φορά η στάση τη απέντη στη Σρι Λάνκα ε, μα βρίσκει σύμφωνο και θεωρώ ότι τιμά επίση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ρίφ, συγγνώμη, τι έχετε να πείτε όμως για την α, Σαουδική Αραβία, όπου έχουμε ακόμα και λιθοβολιδισμούς πολλές φορές εκεί πέρα, ποινές με λιθοβολισμό, Τι έχετε να πείτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί απάντηση. Κοιτάξτε, σαφώς η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με απασχολεί παντού. Δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένε χώρε τις οποίες κατακρίνω και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να επικριθεί για το ζήτημα αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα αναφερθούμε σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη. Είστε προσκεκριμένος να έρθετε εφόσον το επιθυμείτε. Πολύ ωραία. Νομίζω λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ε, βούληση όλων μας είναι, οι νέε αυτές συμφωνίε συμφωνίες θα πρέπει να ασχοληθούν και με προβλήματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο βεβαίως αλλά και με την ε, περισσότερη δημοκρατία στις χώρες αυτές. Αλλά για να απτυχθεί η δημοκρατία αυτή καταλαβαίνετε ότι απαιτείται και οικονομική δραστηριότητα. Πέραν όμω των δικών μας ε, πολιτικών τοποθετήσεων νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε κατά πόσο οι νομικές υπηρεσίες έχουν κάτι να πούν. Γιατί είχαμε ζητήσει συγκεκριμένη γνωμοδότηση από τις νομικές υπηρεσίες. Έχετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συντοποιούμε ότι εδώ πέρα έχουμε μία πρόταση τροποποίησης του κανονισμού, πρόταση που έγινε πριν την έγκριση της συνθήκης της ε, Λισαβόνας και ότι οι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροποποιούνται βέβαια από την έγκριση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Δεν έχουμε εξετάσει ακόμα το ζήτημα πλήρω, Πάντω μπορούμε να το κάνουμε εφόσον το επιθυμείτε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Τόμψον, σας παρακαλώ να είστε πολύ συγκεκριμένος και συνοπτικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Σούλτσα για ε, την ε, πληρέστατη παρουσίαση του, του συστήματος. Δεν χρειάζεται να επανέλθω. Θα ε, είναι λοιπόν πιο σύντομος θα θέλω να, θέλω να μιλήσω λοιπόν για το γεγονός ότι στόχος αυτού του μέτρου είναι να κερδίσουμε χρόνο έτσι ώστε να σεβαστούμε απόλυτα τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου με βάση την, την αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου με βάση τις συνθήκες Λισαβόνας. Δύο σχόλια θα ήθελα να κάνω ε, όσον αφορά την παρέμβαση του κυρίου Σούλτ. Πρώτα απ' όλα είπατε ε, ε, παράταση για τέσσερα χρόνια. Ναι, αυτό νομίζω είπε. Όχι. Αν συμφωνήσουμε στις, ε, στη συνολική αναθεώρηση προηγουμένως δεν πρόκειται να έχουμε τόσο χρονικό διάστημα. Βλέπετε την προσεκτική διατύπωση. Όταν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ε, συναποφασίσει για τις επόμενες ρυθμίσεις. Προφανώς θα μπορούσαν να αρχίσουν να ισχύουν πολύ νωρίτερα. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να δώσουμε περιθώριο για να διονύσετε. Τώρα γιατί καθυστερήσαμε. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ έχουμε νομικές ε, υποχρεώσεις για δημόσια διαβούλευση, για αξιολόγηση αντικτύπου και για τη χρησιμοποίηση των πλέον πρόσφατων στατιστικών για τις γενικευμένες προτιμήσεις που ήταν διαθέσιμα μόλις τον Ιούλιο 2010. Ε, κάναμε τη δημόσια διαβούλευση και απαντώ στο ερώτημα του κ. Σούλτ και το, θέμα, το θέμα αυτό. Δημοσίευση έγινε στις 6 Ιουνίου. Όσον αφορά ε, την αξιολόγηση αντίκτυπου, αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή που βεβαίω ε, θα, θα δημοσιευτεί συνέχεια. Έχουμε ορισμένο βήματα να ολοκληρώσουμε, αλλά ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει με κάτι το οποίο ελπίζουμε να είναι μια συνολική άποψη των πραγμάτων. Άρα λοιπόν, όπως αναφέρθηκε από ένα ή δύο μέλη, οποιασδήποτε ε, προσαρμογές στην τρέχουσα πρόταση θα, γίνουν, ε, θα, θα γινόταν χωρίς αυτή τη συνολική άποψη και αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει. Εμείς εδώ έχουμε μια απλοποιημένη πρόταση, κάνουμε τις ελάχιστες απαραίτητες τεχνικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με θέματα όπως ο κατάλογος διαβάθμιση, την επιλεξιμότητα ε, των, ε, των σημερινών δικαιούχων, το να μπορέσουν και νέες χώρες να υποβάλουν αίτηση. Δηλαδή, κρατήσαμε τις αλλαγές στο ελάχιστο δυνατό για να ε, μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε μία πλήρη συζήτηση για ε, τις ε, επόμενες ρυθμίσεις. Ο κανόνας καταγωγής αφορά κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μέρος μια συνολική πρόταση για το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων. Έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε από τι υπηρεσίε που μα βοηθούν, ε, θα έχει ολοκληρωθεί σύντομα και από του χρόνου θα αρχίσει να εφαρμόζεται, αν είμαστε τυχεροί. Για το θέμα του Πακιστάν. Δεν θα απαντήσω σε λεπτομέρειε. Το μόνο που θέλω να σα πω είναι ότι πιστεύω ότι αποφασίστηκε στη τελευταία ανάλυση ότι εάν, ε, δεν πρέπει τώρα να ανοίξουμε το δρόμο για πιθανές συζητήσεις και για άλλα ζητήματα και ακούσαμε και σήμερα το πρωί χώρες υψηλού εισοδήματος, οι λεγόμενες ε, ε, BRICS που είναι οι χώρες μεσαίου εισοδήματος, θέματα που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας κτλ. κτλ. Οπότε αν ανοίξουμε την πόρτα σε ένα από τα συγκεκριμένα στοιχεία, καταλαβαίνετε ότι το παράθυρο μάλλον τότε ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα στα πάντα. Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε το θέμα του Πακιστάν, και ξέρω και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε κάποια συγκεκριμένη εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα μα απασχολεί το θέμα και ξέρω ότι ο συνάδελφο ε, που θα με διαδεχθεί θα ασχοληθεί με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και ελπίζω να έχει περισσότερε πληροφορίε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Να σταματήσω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, σα ευχαριστώ. Να δώσω λοιπόν πάλι το λόγο στον κύριο Σούλτ. Σα παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομο γιατί έχουμε ξεπλήσει το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίφαση στη συζήτηση αυτή. Αντιθέτως, θεωρώ ότι όλοι κατανοούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ταχύτατη λύση σε ό,τι αφορά το θέμα του rollover, αλλά θα ήθελα να θέσω τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε αυτό ήταν ο σκοπός μου. Γι' αυτό λοιπόν όλοι θα πρέπει να έχουμε κατά νου κατά την επεξεργασία της έκθεσης και καλό και τους κοιόδης εισηγητές να συνεργαστούν προκειμένου να βρούμε μία λύση η οποία θα δώσει μία απάντηση προς όφελος και των εμπορικών σχέσεων στα πλαίσια του GSP, GSP+, αλλά και για να βρεθεί λύση για χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση όπως το Πακιστάν. Ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, ε, σας ευχαριστώ όλους ε, για τις παρεμβάσεις σας. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό και τώρα έχουμε μια συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών. Γι' αυτό σας παρακαλώ όλους όσους δεν ε, ανήκουν στην Επιτροπή μας να αποχωρήσετε. Σας υπενθυμίζω ότι στις συνεδρίες των κεκλειμένων θυρών μπορούν να παραβρεθούν μόνο τα μέλη της Επιτροπής, η Γραμματεία, ε, η εκπρόσωπη των πολιτικών ομάδων, η βοηθή ε, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, ε, ε, της υπηρεσίας των νομικών θεμάτων. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν να φύγετε οι υπόλοιποι από την αίθουσα. Όσοι δεν, έχουν, δεν πρέπει να παραβρεθούν, σας παρακαλώ να φύγετε και ε, θα προβλέψουμε ένα λεπτό για να πάρουμε θέσεις.